We start the meeting. Αρχίζουμε τη συνεδρίαση, λέει η πρόεδρος. Έχετε κάτι να παρατηρήσετε για την ημερησία διάταξη. Όχι. Άρα, εγκρίνεται ω έχει. Θα έχουμε δερμηνία από όλε τι γλώσσε, εκτός από φιλαδικά, κροατικά και μαλτέζικα. Έχουμε ένα νέο μέλος στην Επιτροπή μας ο κ. Ιωακήμ Σταρμπάτη. Έγινε αναπληρωτής στην Επιτροπή Απασχόλησης και εκπροσωπεί την ομάδα ECR. Σημείο με μέσα στις Ανταλλαγή απόψεων με την ετήσια έρευνα για την ανάπτυξη. Αυτό θα γίνει την παρουσία Τάισιν Μοσκοβιζή των Επιτρόπων και του Πρόσχης. Αυτή η συνάντηση θα γίνει αύριο. Και θα ήθελα να έχετε υπόψη ότι θα ξεκινήσουμε στις 8 η ώρα αύριο το πρωί. Πιστεύω θα πάτε για ύπνο νωρί απόψε, ούτως ώστε να μπορέσετε να είσαστε εδώ στις 8 η ώρα. Θα τελειώσετε στις 10. Όχι όμως σε αυτή την αίθουσα. Στο κτίριο Γιάνν στο 4Q2. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή την κοινή συνεδρίαση με την Οικονομική Επιτροπή. Άρα να του δώσετε προτεραιότητα. Στις 3 και 4 με 4 γιατί εδώ θα έχουμε μια άλλη συνάντηση. είναι συνάντηση για το I. Αυτό αποτελεί τη συνέχεια των ε, συζητήσεων, των επαφών που είχαμε και καλέσαμε διάφορους νέους από διάφορα κράτη-μέλη πριν τις ευρωεκλογέ. Επανερχόμαστε τώρα με αυτή την ακρόαση ε, high speed και θα έχουμε και κάποιο κοκτέιλ όπου θα συμμετάσχουν περίπου 100 νέοι. Αυτοί θα παρακολουθήσουν την ακρόαση από εμάς. Έτσι θα δείξουμε στους ε, νέους της Ευρώπης ότι λαμβάνει υπόψη αυτά τα οποία τους απασχολούν στα σοβαρά. Οπότε ελπίζω ότι πολλοί από εσά θα έρθουν να παρακολουθήσουν την ακρόαση iSpeed. Έχουμε επίση ομάδες ε, επισκέψεων είναι 20 επισκέπτες από την Ελλάδα. Κατά τη συνεδρίασή μας επίσης έχουμε κάποιους συνδικαλιστές υψηλού επίπεδου από κάποιο συνδικάτο. Τους έχουμε προσκαλέσει. Όλοι καλοδεχούμενοι. Αύριο επίσης θα έχουμε άλλες δύο ομάδες, το σύνολο 35 πρόσωπα και αυτή η καλοδεχούμενη αύριο. Αν δεν υπάρχει κάποια ένσταση, θεωρώ ότι τα πρακτικά εγκρίνονται. Από την συνεδρίαση της 20ης ενδεκάτου. Εγκρίνονται όσοι έχουν. Υπάρχει κάποια ένσταση, όχι. Πάμε τώρα στο σημείο περιθμών 4 της Μεσής που είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Μόρταν Κέρον που είναι ο Διευθυντής της Υπηρεσίας για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα. Όπως γνωρίζετε πρόκειται για μια υπηρεσία η οποία έχει αναπτύξει ευρύ δραστηριότητα όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα των αναπήρων. τα δικαιώματα των ανηλίκων, των Ρωμά κλπ. Καλώς ορίσατε κύριε Κέρο. Με μεγάλο ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε όσο έχετε να μας πείτε. Thank you very much. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να έχουμε αυτήν την ανταλλαγή. Νομίζω ότι είναι μια μέρα ξεχωριστή. Σήμερα γιορτάζουμε μια πενταετία από την έγκριση της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το γεγονός ότι έγινε νομικός δεσμευτική σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό από μόνο του είναι ένα ορόσημο στην ιστορία των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Ευχαριστώ λοιπόν που με προσκαλέσατε τη συγκεκριμένη μέρα. Και να μην ξεχνάμε ότι η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αφορά και τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα που είναι σημαντικά για την Επιτροπή σας ούτως ή άλλως. Ας δούμε τι έγινε την τελευταία πενταετία και πάμε στην 1η Δεκεμβρίου του 2009 και δούμε το διάστημα σήμερα. Νομίζω ότι είναι πολύ οι λόγοι να είμαστε υπερήφανοι. Πολλά έχουν γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του πλαισίου προστασίας τους Όλοι έχουν αναλάβει διαφορετικά τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους πολίτες. Δεν ανάγκη να τα απαριθμίσω, αλλά νόμοι και πολιτικές που προωθούν την ισότητα, που προστατεύουν τα θύματα, η οδηγία για την προστασία των θυμάτων. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προόδου που βελτιώνει την πρόσβαση στο δικαστικό σύστημα. Με τη νέα Επιτροπή Έχουμε και έναν αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ασχολείται με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό αποτελεί μέρο του τίτλου του ήδη. Και έχουμε και ένα ισχυρότερο Ευρωκοινοβούλιο που πάντοτε προασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα πράγματα λοιπόν έχουν προχωρήσει. Έχουμε ένα πιο σταθερό πλαίσιο. Ταυτόχρονα ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να ε, παραμένουμε σε αυτά που μόλις έχουν γίνει και να αναπαυόμαστε στις δάφνες μας. Υπάρχουν ακόμη πολλές ανάγκες, κυρίως σε σχέση με την οικονομική κρίση. Εάν δούμε κάποιες από τις πολιτικές που γκρίθηκαν εξαιτία της οικονομικής κατάστασης, πολλές από αυτές προκάλεσαν τριγμούς και σε θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, η πρόσβαση στην εργασία, το δικαίωμα εργασίας και η ελευθερία ή η απαλλαγή από ε, συμπεριφορές διακριτικής μεταχείρισης. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω το παράθεμα του Πάπα Φραγκίσκου όταν ήρθε στο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα. Απλώς ένα πράγμα θα πω. Τι αξιοπρέπεια να έχει ένας άνθρωπος όταν πρέπει να υποστεί κάθε είδους διακριτική μεταχείριση. Τι αξιοπρέπεια μπορεί να βρει εάν εκείνη ή εκείνος δεν έχει τρόφιμα ή τα βασικά προς επιβίωση. Ακόμα χειρότερα όταν δεν έχει δουλειά, δουλειά η οποία ακριβώς αυτή προσδίδει την αξιοπρέπεια στον άνθρωπο. Αυτά είπε και νομίζω ότι αυτά βρισκόνται στην καρδιά των ενδιαφερόντων της Επιτροπής σας. Αλλά και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να προσπαθήσω λίγο να παρουσιάσω το τι κάνει ο Οργανισμός των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τονίζοντας ε, και παίρνοντα ω παράδειγμα τρει ευάλωτε ομάδε του πληθυσμού τι σημερινέ συνθήκε, του ανθρώπου με αναπηρίε, του Ρωμά και τα παιδιά. Εάν κοιτάξετε του ε, ανθρώπου με αναπηρίε, θα το γνωρίζετε εσεί, είναι πολύ ψηλό το ποσοστό αυτών των ανθρώπων που είναι άνεργοι. Πολύ μικρό μέρος των ανθρώπων αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δουλειά και φτάνουμε περίπου στο 70% το συγκρίνουμε με το συνολικό ενεργό πληθυσμό. Είναι τεράστια η διαφορά μεταξύ των ανθρώπων που έχουν ε, αναπηρίες και αυτών που δεν έχουν. Κάτι παρόμοιο ισχύει και για την εκπαίδευση. Στα ανώτατα επίπεδα, στην εγκατάλειψη του σχολικού συστήματος, πολλοί είναι αυτοί από τους ανθρώπους με αναπηρίες που δεν ολοκληρώνουν τον εκπαιδευτικό κύκλο και φτάνουμε έτσι στην ένδια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Περνάει κανείς σε έναν φαύλο κύκλο εφόσον ανήκει σε αυτή την ομάδα. Γι' αυτό η σύμβαση του ΟΗΕ για, την, ε, για, για τους ανθρώπους με αναπηρίες, η CIPD, είναι ένα ορόσημο. Είναι μια απόπειρα από την πλευρά της διεθνούς κοινότητας να αντιστρέψει αυτή την αρνητική τάση. Μια τάση στην οποία δεν είναι μόνη της η Ευρώπη. Και δεν είναι μοναδική για την Ευρώπη, διότι παρόλα αυτά η Ευρώπη πρώτη φορά κυρώνει μια τέτοια παγκόσμια σύμβαση. Αυτό έχει και συνέπειες για την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Πρώτα απ' όλα η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και ο ίδιος οργανισμός μου θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις επιταγές της ε, σύμβασης. Κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και κάνουμε μια συντονισμένη, έχουμε συντονισμένες ενέργειες για να λειτουργήσουν όλα αυτά πιο εύρυθμα. Όμως η αρμοδιότητα της Ένωσης ως προς τα κράτη-μέλη ε, για τα θέματα αυτά είναι αρμοδιότητα που υπερισχύει σε ό,τι αφορά την ίδια κρατική μεταχείριση και την εργασία. Αυτοί είναι δύο βασικοί τομεί. Οι νέοι κανόνε για τα διευθυντικά ταμεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ ισχυροί. Προβλέπουν για τι ομάδε των ανθρώπων με αναπηρίε να <clears throat> συμμετέχουν σε διαβουλεύσει και να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκε του κατά, ε, κατά τον σχεδιασμό νέων προγραμμάτων. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα και βλέπουμε πάλι τη σημασία του να υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο έχει θεσπιστεί ακριβώ μέσω τη σύμβαση. Έπειτα ως προς το ίδιο θέμα να τονίσω ότι θα καλωσορίσουμε ένα ακόμη ισχυρότερο πλαίσιο παρακολούθησης για να μπορεί το Κοινοβούλιο μαζί με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων την Επιτροπή και το κίνημα για του ανθρώπου με αναπηρίες να ε, μελετήσουμε τελεχώ τα θέματα αυτά, να καταρτήσουμε ένα πρόγραμμα δράση που να καλύπτει τις βασικές μέρημνες σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά όργανα αλλά και όπου αλλού έχουμε μια μεικτή αρμοδιότητα. Ο Οργανισμό των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων έχει εργαστεί για τα θέματα των αναπηριών των προσώπων με αναπηρίε επί πολλά χρόνια, ιδίω για την ανεξάρτητη ζωή, την αυτονόμηση των προσώπων αυτών, που είναι πρώτη προτεραιότητα. Θα θέλαμε να τα ξαναδούμε μαζί σας όταν προχωρήσουμε. Να στραφώ τώρα στην άλλη ομάδα που ήθελα να σχολιάσω. Στα θέματα των Ρωμά. Εδώ ο Οργανισμό των Θεμελιωτών Δικαιωμάτων έχει αναλάβει, έχει μάλλον διεξαγάγει την πλέον σφαιρική μελέτη που έχει γίνει ποτέ στην Ευρώπη ή οπουδήποτε αλλού. μιλήσαμε με 800.000 μέλη νοικοκυριών Ρωμά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, κατά πρόσωπο διαζώσει για θέματα διακριτική μεταχείριση, κοινωνικού αποκλεισμού και άλλα βασικά θέματα για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αλλά πέραν από αυτού ε, μιλήσαμε περίπου με 20.000 ε, ανθρώπου που είναι απλώς γειτονέ τους για να δούμε γενικότερα τα θέματα φτώχεια στι συγκεκριμένες περιοχές των κρατών μελών και να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τους Ρωμά και επίση ήρθαμε σε επαφή και με 300 ε, δήμου και κοινότητε, ε, φορεί τοπική αυτοδιοίκηση, για να δούμε πώ ασχολούνται με τα θέματα αυτά σε καθημερινή βάση. Όλα αυτά τα δεδομένα μπορείτε να τα δείτε και στον ιστότοπό μα. Ε, αν τα διαβάσετε, είναι πραγματικά σοκαριστικά. Αλλά ένα-δυο σχόλιο μόνο ε, από πλευρά μου. Πρώτον, ο αναλφαβητισμό. 15% των Ρωμά, των ανδρών και περίπου 25% των γυναικών δεν μπορούν να διαβάσουν ή να γράψουν. Εάν το συγκρίνουμε με το τι συμβαίνει στους γειτονές τους, όχι το γενικότερο πληθυσμό, απλώς όσους μένουν δίπλα τους, είναι περίπου 1% ε, ο αναλφαβητισμός στον γενικότερο πληθυσμό. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Και αυτό φαίνεται εάν δει κανείς και την ε, συστηματική παρακολούθηση του σχολείου, την εγκατάλειψη του σχολικού συστήματος που είναι πολύ μεγαλύτερη στους Ρωμά από ό,τι στους γειτονές τους. Αυτό έχει ένα αντίκτυπο, όπως θα περιμένατε, και στα ποσοστά ανεργίας. Τριπλάσια ανεργία στους Ρωμά από ό,τι στους υπολείπους. Στους γειτονές τους συγκεκριμένα. Είναι λοιπόν μεγάλη αυτή η πρόκληση. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να ε, βεβαιωθούμε ότι τα κράτη-μέλη θα συνεχίσουν να εργάζονται προκειμένου οι στρατηγικέ ένταξει των Ρωμά θα αποδώσουν καρπούς. Αυτές οι στρατηγικέ είναι πολύ σημαντικές κινητήριε δυνάμεις για αλλαγή. Η αλλαγή αυτή χρειάζεται στα κράτη-μέλη. Χρειάζεται στα κράτη-μέλη όπου υπάρχουν μεγάλε κοινότητε Ρωμά. Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα συνεχίσει την ε, μελέτη αυτού του τύπου ε, σε επαφή με τον πληθυσμό των Ρώμα, σε πολλά και βεβαίως έχουμε και μια ομάδα εργασία όπου συγκεντρώνονται μέλη από όλα τα κράτη-μέλη για να δούμε πώς μπορούμε καλύτερα να παρακολουθήσουμε την πρόοδο στην, ε, στο επίπεδο της ένταξης των Ρώμα. Θέλουμε δηλαδή ένα υψηλότερο επίπεδο λογοδοσίας για το πώς χρησιμοποιούνται τα ε, κρατικά αλλά και ευρωπαϊκά κονδύλια. Είναι λίγοι οι πόροι εδώ, αλλά πρέπει να αξιοποιούνται όσο το δυνατόν καλύτερα. Τέλος, για τα παιδιά. Έθιξα ήδη το θέμα των Ρωμά και των παιδιών τους μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος. Εάν δείτε τώρα το γενικό πληθυσμό των παιδιών, βλέπουμε ότι τα παιδιά έχουν πληγεί ιδιαίτερως από την οικονομική κρίση. 30% ε, των παιδιών βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχεια ή κοινωνικού αποκλεισμού. Δραματικά τα στοιχεία. Πρέπει να προσέξουμε στην Ευρώπη να μην χάσουμε μια ολόκληρη γενιά μέσα από τα χέρια μα. Για αυτό το λόγο ο Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και πάλι εργάζεται σκληρά και σε αυτόν τον τομέα. Σε αυτή, τη στιγμή, σε αυτή τη φάση κοιτάζουμε το τι γίνεται με τα θέματα βίας ή κακοποίησης παιδιών με αναπηρίες αλλά και την, τα συστήματα προστασίας των παιδιών γενικότερα. Πώς προστατεύουν ε, τα κράτη-μέλη τα παιδιά, πώς ε, ρυθμίζουν την πρόσβασή τους στο δικαστικό σύστημα και τη δικαιοσύνη. Αυτά είναι ορισμένα από τα βασικά θέματα που μας απασχολούν, με τα οποία ήθελα να σας απεικονίσω πώς εργαζόμαστε στον οργανισμό. Απλώς να ολοκληρώσω, ε, τονίζοντας κάποια ακόμη στοιχεία για την επόμενη χρονιά. Αυτά που επίκυνται. Η πρώτη έκθεση που θα δημοσιεύσουμε θα αφορά ιδιαίτερω και τη δική σας τη δουλειά. Μια έκθεση για την ακραία εκμετάλλευση στην Ευρώπη. Δηλαδή την σύγχρονη, όπως θα την έλεγα, δουλεία. Δεν είναι το φαινόμενο απαράλλαχτο σε σχέση με το παρελθόν. Έχει πάρει άλλη μορφή, αλλά μιλάμε πραγματικά για δουλεία στην Ευρώπη. Υπάρχει αυτό και από νομική σκοπιά, αν το δει και από κοινωνική. Μιλήσαμε με εργαζομένους και επιθεωρητές εργασίας για να δούμε πού εντοπίζονται οι αδυναμίες σήμερα στην Ευρώπη. Μια άλλη έκθεση που θα ακολουθήσει στις αρχές του 2016 θα είναι μια έκθεση η συνέχεια της πρώτης μελέτης που είχαμε κάνει για τις εθνοτικές μειονότητες τότε είχαμε μιλήσει με 25.000 ε, μέλη εθνοτικών μειονοτήτων και αυτό θα επαναληφθεί. Είναι η πρώτη μελέτη που ε, συνεχίζεται που έχει και δεύτερο σκέλος και θα μας δείξει πώς εξελίσσονται οι διάφορες τάσεις που τότε έχουμε παρατηρήσει. Υπάρχει οπισθοδρόμηση, υπάρχει πρόοδος, θέλουμε να δούμε τι γίνει σφαιρικότερη εικόνα και είναι μια νέα διάσταση στις μελέτες που έχουμε κάνει ως τώρα αυτή θα δούμε πώς οι εθνικές μειονότητες και άλλες μειονότητες οδεύουν προς τους στόχους το 2020, όπως τους είχαμε καθορίσει πριν από κάποια χρόνια. Κινώντας τη σωστή κατεύθυνση. Θέλουμε να δούμε τι πορίσματα υπάρχουν και να τα συζητήσουμε μαζί σας. Εν είδη συμπεράσματος, λοιπόν, επικεντρωνόμαστε στους φραγμούς που υπάρχουν για να γίνει κοινωνία πραγματικά συμμετοχική. Εμπόδια που σχετίζονται με διακριτική μεταχείριση στην αγορά εργασία, το εκπαιδευτικό σύστημα και άλλου ζωτικού τομεί. Εδώ έχω μία μικρή παράκληση προς εσάς. Βοηθήστε μας, ασκώντας πίεση όπως κάναμε ήδη από το 2008, να επιτελεστεί πρόοδος για την οριζόντια οδηγία τη Ευρωπαϊκής Ένωση και για την κριτική μεταχείριση. Για όσου είναι θύματα κοινωνικού αποκλεισμού στις ευρωπαϊκές κοινωνίες η οδηγία αυτή θα κάνει τεράστια διαφορά. Είναι σημαντική και χαίρομαι που ήδη έχει περάσει και είναι μια από τι πρώτε προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήδη έχουμε μια πενταετία νομική ισχύω τη χάρτα. Κατά την άποψή μου, υπάρχει ένα τομέα, αυτό των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών, όπου θα μπορούσε να έχει υπάρξει μεγαλύτερη πρόοδο. Θα ήθελε μελέτη αντικτύπου για τα θεμελιώδη δικαιώματα να είναι πιο ε, καλά θεμελιωμένη στο μέλλον, πιο καλά τεκμηριωμένη. Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών. Δεν μιλάμε για πυρηνική φυσική, μιλάμε για κάτι που μπορεί να γίνει, είναι εφικτό και θα έχει έναν σημαντικότατο αντίκτυπο. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Thank you. Now ε, σας ευχαριστώ. Και τώρα, ποιος θέλει τον ε, λόγο από το Ευρωπαϊκό Κόμμα. Πρώτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Διευθυντά για το τοπίο το οποίο μας περιγράψατε με τόσο πλήρη τρόπο για ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει τόσο πολύ ε, ε, και, και τον καθένα από εμά χωριστά, αλλά και όλου μαζί όσον αφορά την ε, αποτροπή μα για την απασχόληση κοινωνικέ υποθέσει. Εγώ τώρα θέλω να επανέλθω σε κάτι που είπατε στο συμπέρασμά σα, ότι έχουμε κάνει βήματα πρόοδο, αλλά βεβαίω και ε, την τελευταία πενταετία βεβαίω και κάναμε κάποια πρόεδρο. Όταν όμω αντιμετωπίζω την πραγματικότητα όσον αφορά την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίω όσον αφορά τις ε, μειονότητες αναρωτιέμαι μήπως πρέπει για πρώτη φορά να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια στην διοίκηση ώστε να κινητοποιηθούν ε, στα κράτη-μέλη η διοίκηση, η διοικήσεις τέλο πάντων για προς εκείνη την κατεύθυνση και όσον ε, μας είπατε ότι έχουμε αυτή την γενική σύμβαση η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί, θα πρέπει να τήρηθει και βασικό σημείο που ορίζεται εκεί και θα πρέπει να γίνει σεβαστό από την διοίκηση ε, είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει από τα κράτη-μέλη. Για πετε μας, έχετε κάποιο είδους ε, ε, αντίληψη πιο συγκεκριμένη όσον αφορά τις προόδους που έχουν σημειωθεί ίσως κάπως αισιόδοξα, ίσως και για το την πορεία που έχουμε ακόμα μπροστά μας πρέπει να την κάνουμε ε, σαν ρεαλιστές ούτως ώστε να δούμε ε, με τι τρόπο εσείς θεωρείτε ότι μπορούμε να ε, προωθήσουμε το, το έργο της διοίκησης για το ζήτημα αυτό. Κατά δεύτερο, μας αναφέρατε τους ανηλίκους για τον κίνδυνο από τη φτώχεια. Είδατε και το σχολείο είναι ένα βασικό εργαλείο κοινωνικής ένταξης για αυτούς τους νέους. Έχετε κάποια άποψη το τι γίνεται στα επιμέρους κράτη-μέλη ε, όσον αφορά κάποιες αξιόλογες πρακτικές και συγκεκριμένα το τι ισχύει όσον αφορά την ε, εκπαίδευση από απόσταση. Να δούμε δηλαδή μήπως αυτοί οι ανήλικοι μετανάστες, αυτοί οι νέοι ε, τι κάνουν. Τρίτη μου ερώτηση, πάντα στο πνεύμα μιας ρεαλιστικής αντιμετώπισης κύριε Διευθυντά, ακριβώς πού βρίσκονται τα αδύνατα σημεία. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κρίστενσεν από τους Σοσιαλιστές. Σας ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσω και εγώ για την παρουσίασή σας. Και φυσικά δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τις προτεραιότητες. Θα πρέπει να κάνουμε πιο πολλά για τους ανάπηρους, για τους τρομά και για τα παιδιά. Κοιτώντας ε, τον κόσμο στην Ευρώπη, η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων είναι πάρα πολύ σημαντικό δικαίωμα και επίτευγμα, αλλά ακόμα και πολλές δυσάρεστες ε, περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει αξιοπρεπής ε, μεταχείριση του ατόμου. Οι προθέσεις πίσω από τους νόμους ε, στην Ευρώπη, το γεγονός δηλαδή ότι το όταν πηγαίνουμε σε, μια κράτη, σε ένα άλλο κράτος μέλος πρέπει να ακολουθούμε τους κανόνες. Οι προθέσεις λοιπόν είναι αναμφίβολα σωστές, αλλά δυστυχώς εφαρμόζονται με λάθος τρόπο και τελικά υπάρχει διακριτική μεταχείριση και σε ό,τι αφορά τις μισθολογικές ε, κλίμακες. Έχετε κάποια ιδέα για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στην Ευρώπη? Η κυρία Στάινρουκ από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων υποθέτω ότι έχει πάρα πολλή δουλειά μπροστά του ακόμα. Δύο ερωτήσει έχω να σα θέσω. Στι 3 του έχουμε την Διεθνή ημέρα για τα άτομα με αναπηρία. Η συμμετοχή των ΑΜΕΑ στην αγορά εργασία και η πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι κάτι το οποίο δεν έχει με το έχουμε εξασφαλίσει σε όλες τις περιπτώσεις. Έχετε κάνει μελέτες εσείς για το πώς διαμορφώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο η κατάσταση. Και κατά δεύτερον, ε, στην ε, αγορά εργασίας στην Ευρώπη έχουμε διάφορες εξελίξεις και ο κύριος Κρίστανσεν ήταν υπεύθυνο για ήταν ε, εισηγητής για μια έκθεση για τις νέες μορφές εργασίας άτομα τα οποία έχουν θέση εργασίας αλλά δεν μπορούν και εξαρτώνται από τα κοινωνικά ε, επιδόματα για να επιζήσουν. Από την άλλη, διάφορες άλλες νέες μορφές συμβάσεων, όπως ε, συμβάσεις ε, κοινή απασχόλησης σε διάφορους εργοδότες. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε κατά πόσον αυτό είναι αντίθετο και δεν συνάδει με τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Σας ευχαριστώ. Από την ομάδα της Γκούε, η κυρία Κλάρη. σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Κέρομ για τις ε, παρατηρήσεις του, για το εικόνα που σχημάτισε για μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πώς λειτουργεί ο οργανισμός θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σε ό,τι αφορά το θέμα που δείξατε για την σύγχρονη δουλεία 880.000 άτομα εικάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι εργάζονται υπό συνθήκες δουλείας. Πρόκειται για κάτι απαράδεκτο έχει ο οργανισμός μέσα στη διάθεσή του για να καταπολεμήσει την κατάσταση για να εξετάσετε τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον για να καταπολεμήσουμε την κατάσταση αυτή. Έχω την αίσθηση ότι τα πράγματα είναι μάλλον στατικά και δεν εξελίσσονται. Μπορούμε όμως κάτι να κάνουμε. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο κύριος Ηλικιώτης. <laughs> From the Sorry from my pronunciation. Ναι, ε, κύριε Κιάρου, ε, πολύ σωστά αναφερθήκετε στα προβλήματα και στα πορίσματα που ο οργανισμός, ο σας διαπιστώνει ε, και για τα προβλήματα των παιδιών και την παιδική δουλεία. Όμως αυτό που δεν ακούμε είναι και είναι η πηγή αυτών των προβλημάτων. Ιδιαίτερα στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, λόγω της βαθιάς οικονομικής κρίσης, αλλά και των νεοφιλεύθερων πολιτικών λιτότητας που εφαρμόζονται, που επιβάλλονται θα έλεγα από τα μνημόνια και τις τρόικες, παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, των αναπήρων, των συνταξιούχων, θα έλεγα όλων των ευάλωτων ομάδων. Βλέπουμε το κοινωνικό κράτος να συρρυκνώνεται, να δημιουργείται ανισότητα σε με το φύλων, να διευρύνεται ε, η, αυτή η ανισότητα. Ε, παιδιά όπως αναφέρεται να εγκαταλείπουν το εκπαιδευτικό σύστημα, να υπάρχουν σοβαρά ελλείμματα στην ιατροφαρμακευτική ε, περίθαψη ε, παράλληλα σε αυτά τα κρατημέλη βλέπουμε να απορριθμίζεται ε, η εργασία διότι όταν μιλούμε για δήλωτη εργασία είναι γιατί οι εργασιακές σχέσεις ε, ε καταλύονται μέσω αυτών των νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Ε, η ανεργία επίσης κάνει άλματα ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους και ταυτόχρονα είναι και πηγή που ενισχύεται η ξενοφοβία και ο ρατσισμός ακριβώς πέραν από το να αναφέρουμε στοιχεία, ο οργανισμός σας μελετώντας αυτά τα προβλήματα και συγκεκριμένες προτάσεις καταθέτει ε, ε, και σε σχέση ακριβώς ε, με τις πολιτικές αυστηρής λιτότητας που εφαρμόζονται που κατά την άποψή μας είναι και η πηγή όλων αυτών των προβλημάτων που και εσείς διαπιστώνετε κύριε Γκάρου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχουμε άλλους τέσσερις που θέλουν να υποβάλουν ερωτήσεις. Κύριε Λόπες Μπερμπέγιο, πρώτη, από την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά. Σας ευχαριστώ. Πρώτα-πρώτα να σας ευχαριστήσω για όσα έρθετε να μας πείτε. Συμφωνώ με την ανάλυση στην οποία προδίκατε όσον αφορά τη φτώχεια και τα σχετικά. Στην Ισπανία δυστυχώς, λόγω της εφαρμογής των πολιτικών λιτότητας, βρεθήκαμε δεύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την μεγαλύτερη φτώχεια για τους ανηλίκους. Επίσης είχαμε για κοινωνική πολιτική και για πολιτική για τους ηλικιωμένους μεγάλες περικοπές και γενικά για τον κόσμο της δουλειάς περικοπές. Οπότε τελικά υπήρξαν επίσης περικοπές όσον αφορά και τα υγειονομικά για τους μετα, μετανάστες και φυσικά έχουμε έτσι και θέματα δυσμενούς διάκρισης. Συμφωνούμε με όσα είπατε, αλλά δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μια συνταγή για όλους. Θα έπρεπε νομίζω να προσέξουμε ιδιαίτερα κάποιες ομάδες, ας πούμε τις γυναίκες, γιατί Ό,τι αρνητικό υπάρχει, ό,τι, ό,τι, ό,τι ευάλωτο υπάρχει τελικά χτυπάει τις γυναίκες στις ομάδες που αναφερθήκαμε. Ας πούμε στις, στην Ισπανία οι ανάπηρες γυναίκες ε, ε είναι πιο, ε, έχουν, έχουν οκτώ μονάδες παραπάνω από την ανεργία των υπολείπων. Και ήδη οι ανάπηροι έχουν όλοι μαζί 40% περισσότερη ανεργία από όσους έχουν άλλες κοινωνικές ομάδες. Εμείς πάντως υπολογίζουμε στο δικό σας έργο για να διορθώσουμε τα οικοσκήμενα να δούμε πώς θα πετύχουμε τους στόχους ε, για το 2020, για, για την παιδεία, για τη φτώχεια. Πάντως θα πρέπει να προχωρούμε συντονισμένα όσον αφορά αυτούς τους κοινωνικούς στόχους και να δίνουμε τη μάχη μας όποτε η λιτότητα έχει προτεραιότητα εναντί αυτών των, ε, των κοινωνικών στόχων. Ε, ο κ. Φουντούλη για του μη γεγραμμένους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Γιάρου. Ε, έχετε εξετάσει το θέμα της αντιμετώπισης ότι το θέμα της αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας είναι συνδεδεμένο άρρηκτα με το πρόβλημα των παράνομων μεταναστών. Λέω παράνομοι μετανάστες και όχι παράτυποι όπως θέλουν, θέλουν κάποιοι να τους αποκαλούν, γιατί τα κράτη έχουν νόμους που πρέπει να γίνουν σεβαστοί και όχι τύπους. Μην μπερδεύουμε τον ανθρωπισμό με την νομιμότητα κάθε παράνομο μετανάστη, τον οποίο εκμεταλλεύονται κάποιοι λόγω τη ανάγκη του, στερούν θέσει εργασία από του ανέργου που ειδικά στι χώρε όπω είναι η Ελλάδα είναι 1,5 εκατομμύριο. Η αδήλωτη εργασία δεν συνεισφέρει ούτε στα φορολογικά εισοδήματα τη χώρα, ούτε στι ασφαλιστικέ εισφορέ των ταμείων που βρίσκονται στα όρια τη κατάρρευση. Για του Ρωμά, επειδή έχω μιλήσει με πολλού Ρωμά στην Ελλάδα, αναρωτηθήκατε ότι η επιλογή του να είναι στο περιθώριο είναι από δική του πρόθεση. Έχετε εξετάσει το θέμα από την πλευρά του ότι θέλουν να κρατήσουν την αυτοτέλειά τους και ότι δεν θέλουν να ενσωματωθούν στο δικό μας κόσμο. Μήπως οι ίδιοι θέλουν να βρίσκονται στο περιθώριο και όχι να ακολουθούν τους νόμους και τις υποχρεώσεις απέναντι στα κράτη. Ευχαριστώ. Mr. From ECR. Κύριος από τους ε, συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Θα μιλήσω σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει... Είναι πολύ σημαντική η ανάλυση αυτή που μας παρουσιάσατε, αλλά ως κοινωνιολόγος έχω την ε, αίσθηση ναι. ότι μας ε, παρουσιάσατε κλασικά παραδείγματα παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κλασικές ε, ομάδες, Σύντη και Ρώμα, τα... τις οποίες τις ακούμε και στα μέσα ενημέρωσης για τις άλλες ομάδες, για τους ανάπηρους. Ήθελα να ρωτήσω ότι αν ο οργανισμός παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις, όπως για παράδειγμα στη Γερμανία με την εισρωή Ρωμά στην Γερμανία, έγιναν κάποιες ε, πολύ λεπτές μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Μια δεύτερη ερώτηση. Σήμερα αντιμετωπίζουμε μια πιο σύγχρονη και πιο σύνθετη, αν θέλετε, μορφή διακριτικής μεταχείρισης. Πιστεύω, είναι η δική μου η εντύπωση τουλάχιστον αυτή, ότι αυτά που μας αναφέρατε αποτελούν μόνο ένα τμήμα της Ευρώπης. Τι γίνεται με το άλλο πολιτικό τμήμα της Ευρώπης και τι εννοώ. Τα φαινόμενα που τα ανέφεραν οι συνάδελφοι. Η ολική κατάρρευση, για παράδειγμα, του συστήματος προστασίας υγείας της υγειονομικής περιθάλψης. Υπάρχουν χιλιάδες άτομα που έχουν καρκίνο για παράδειγμα και χρειάζεται να, να περιμένουν για τη θεραπεία τους. Κάτι το οποίο στην Πολωνία ονομάζουμε τα ευρωορφανά. Παιδιά που μεγαλώνουν μόνο τους, γιατί οι γονεί του είναι στο εξωτερικό. Η διακριτική μεταχείριση σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των επιχειρήσεων. Τέλος. Αυτό που επίσης παραβιάζεται στην Ευρώπη είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, το δικαίωμα του ψηφίζει. Στην Πολωνία είχαμε σαφείς παραβιάσεις πρόσφατα και από ό,τι ακούω παρόμοια περιστατικά παρουσιάστηκαν και στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία. Η εμπιστοσύνη λοιπόν του κόσμου στους πολιτικούς θεσμούς ε, καταραίει και αυτό επειδή αισθάνεται το άτομο περιθωρεποιημένο. και αυτό αφορά ολόκληρες περιοχές, ολόκληρες περιφέρειες και εκ παραλλήλου λοιπόν παραβιάζονται τα πολιτικά δικαιώματα και αυτό είναι κάτι το οποίο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρέπει να το ξεχνάμε, πρέπει να το σκεφτούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην Ευρώπη, στο σύνολο της Ευρώπης. Δεν αμφισβητώ τη σημασία των προβλημάτων που μας αναφέρατε εσείς, μην με παρανοήσετε. Είναι σαφές ότι υπάρχουν και αυτά τα προβλήματα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να συμπληρωθούν και κάποια άλλα σημεία, όπως αυτά που ανέφερα. Ευχαριστώ, Σάντρα, από την ομάδα του ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για όλα τα ενδιαφέροντα στοιχεία που μας παρουσιάσατε και που μας δείχνουν τι δουλειά έχουμε ακόμη μπροστά μας. Ήθελα να σταθώ σε ένα σημείο πολύ συγκεκριμένο που αφορά τα άτομα με αναπηρίες. Στη Γαλλία, όπως και σε άλλες χώρες φαντάζομαι, αλλά θα μπορείτε εσείς να μου πείτε καλύτερα, οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση ως προς την ε, απασχόληση ανθρώπων με αναπηρίες. Όμως, ας ε, σκεφτούμε ότι συχνά επιχειρήσεις, αντί να προσλάβουν τέτοια άτομα, προτιμούν να πληρώσουν πρόστιμα. Αυτό για διαφορετικούς λόγους, ως επιτοπλίστων εξηγώντα ότι δεν είναι οργανωμένες ως προς την οργάνωση, τέλος πάντων από εργονομική σκοπιά για να υποδεχτούν τέτοια άτομα. Ήθελα να μου πείτε τι συμβαίνει σχετικά στις υπόλοιπες χώρες. Και η Γαλλία είναι ένα από τα παραδείγματα. Για να σταθώ σε αυτό έχουμε ένα νομικό ένα νομοσχέδιο που θα έπρεπε να εφαρμόζεται για την πρόσβαση του κοινού, αλλά θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στον χώρο των επιχειρήσεων. Υπάρχει, υπάρχει τέτοιο νόμο, αλλά ε, στην πράξη δεν εφαρμόζεται. Παρακαλώ λοιπόν να μα πείτε εσεί για τι υπόλοιπε χώρε. Ο κύριος ε, Μαρτέν από τους μη γεγραμμένους. Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε, μα μιλήσατε για τα άτομα με αναπηρίε, τα παιδιά και του Ρωμά και για το πρόβλημα τη παιδική δουλεία στην Ευρώπη. Βεβαίω, ε, τα άτομα με αναπηρίε είναι ε, το πλέον ευάλωτο τμήμα του πληθυσμού μεταξύ των συμπολιτών μα. Και παιδιά και ηλικιωμένοι και ανάπηροι ε, χρειάζονται σαφώ στήριξη. Ω προ του Ρωμά, είπατε ότι πρέπει οπωσδήποτε να προσπαθήσουμε να του εντάξουμε. Ναι, γιατί όχι. Όμως εγώ σας θέλω το εξή ερώτημα. Οι Ρωμά θέλουν οι ίδιοι να ενταχθούν. Για να ξεκινήσουμε από αυτό το πρώτο πρόβλημα και όταν θα αποφασίσουν εκείνοι να ενταχθούν, ε, και δεν μου αρέσει και ο όρος ένταξη, δεν τον ε, εκτιμώ ιδιαίτερα, προτιμώ τον όρο αφομοίωση. Εκεί θα μπορούσαμε ίσως να τους διευκολύνουμε, ως προς τα παιδιά. Ναι, ωραία τα λέτε, αλλά η Ευρώπη πώς θα μπορούσε να υποκαταστήσει τις ομάδες των γονέων, το ρόλο των γονέων τον ίδιο. Αυτοί δεν πρέπει να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους, να τους δώσουν αγωγή και εκπαίδευση. Ε, πρέπει λοιπόν ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Διευθυντά να σκεφτούμε πρώτα απ' όλα τι κάνουν οι γονείς που εγκαταλείπουν τα παιδιά τους. Αυτό αφορά και τον αναλφαβητισμό και το εκπαιδευτικό σύστημα και όλα τα υπόλοιπα και ως προς την δουλεία στην Ευρώπη. Θίξατε το φαινόμενο της δουλείας στην Ευρώπη, νεοαπικιοκρατικές τάσεις του κόσμου μας. Αλλά για να το δούμε καλύτερα. Η Ευρώπη δεν φταίει που έχει καταστήσει καινού νοήματο το Σέγγεν με την απελευθέρωση της κυκλοφορία των ε, ε, αγαθών, των υπηρεσιών και κυρίω των προσώπων. Η ίδια δεν προέβλεψε την οδηγία για του εργαζομένου σε απόσπαση. Η ίδια δεν έχει πλέον καταργήσει τα σύνορα γύρω τη Μήπως κάνοντας όλες αυτές τις κινήσεις η Ευρώπη άφησε κάποιους πονηρούς να αναλάβουν δράση δουλεμπόρου ε, όπως στη Μεσόγειο. ή το να προσφέρουν στέγη σε μετανάστε φορές χάνουν τη ζωή τους λόγω πυρκαγιάς ή στο δεύτερο και τρίτο υπόγειο δουλεύουν για εξευτελιστικές τιμές. Αυτά ίσως να είναι οι λόγοι που οδήγησαν στην ε, σύγχρονη δουλεία να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε του αλλοδαπού που έρχονται, όπω είπατε. Θετική διακριτική μεταχείριση όμω λέγεται αυτό. Και ε, εδώ και 20 χρόνια αυτό προωθούν τα 28 κατημέλη. Αλλά καλά είναι να γνωρίζετε και φαντάζομαι το ξέρετε γιατί από τη δουλειά σα την καθημερινή. Η θετική αυτή διακριτική μεταχείριση έχει καταλήξει στην προτίμηση των ξένων τελικά. Δηλαδή πολλές φορές τα κράτη-μέλη, τα εθνικά κράτη ε, δίνουν προτεραιότητα στους ε, αλλοδαπούς και όχι στους δικούς τους πολίτες. Φοβούμε λοιπόν ε, κύριε Διευθυντά και με όλο το σεβασμό στο έργο σας ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα που ευαγγελίζεστε τελικά έχουν γίνει τα δικαιώματα των ξένων. Okay, 10 minutes for you to Τώρα λοιπόν έχετε δέκα λεπτά κύριε για να απαντήσετε όλες αυτές τις ερωτήσεις. But I'm you can make it. Είμαι σίγουρη όμως ότι θα τα καταφέρετε. Ναι, ναι, είστε διευθυντής. Εμείς θα πρέπει να τα απαντάμε τα ερωτήματα. Εσείς, όχι υποχρεωτικά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες αυτές τις μεστές ερωτήσεις, τις ε, εύστοχες. Δύσκολα ε, σε 10 λεπτά θα έπρεπε κάθε ερώτημα να απαντάτε με ένα ολόκληρο σεμινάριο που τέλος πάντων θα προσπαθήσω. Η πρώτη ερώτηση του κύριε Σωτό. Όσον αφορά τις μειότητες στην Ευρώπη και τη διοίκηση, τι γίνεται σε τοπικό, σε εθνικό επίπεδο. Ρωτήσατε αυτό, εάν κατάλαβα καλά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί αν ρίξουμε μια ματιά στο τι γίνεται με τα θεμελιώδη δικαιώματα, είπαμε τι γίνεται με για ανάπηρο, Ρωμά. Πολλέ φορές αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα ε, και οι παραβιάσει τους γίνονται γιατί το σύστημα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα φαινόμενα σε επίπεδο δημοτικό, περιφερειακό, ακόμα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλώς δεν μπορούμε να έχουμε μια κοινή προσέγγιση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά από αυτά τα προβλήματα. Θα σημειώνουμε μεγάλη πρόοδο εάν υπήρχε περισσότερη συνεργασία, οριζόντια αντιμετώπιση μεταξύ των διάφορων εμπλεκομένων και όχι αντιμετώπιση κάθετη του ΣΥΠΗ μεταξύ των διαφορετικών επίπεδων. είπαμε για 21 Δήμους και με το που έγινε αυτή η συνεργασία και η συνεργασία διαφόρων φορέων να δούμε τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε. Και μιλάμε τώρα για το τι γίνεται και για τους Ρωμά και για τον υπόλοιπο πληθυσμό. Τι γίνεται με τους ε, αναπήρους, με τις εθνικές, εθνοτικές μειονότητες και τις άλλες μειονεκτούσες ομάδες. Κάθε φορά υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση βέβαια, αλλά υπάρχουν περίπου κοινά προβλήματα πολλά. Ας πούμε, τι γίνεται με τους Ρωμά και τις εθνικές στρατηγικές. Κάποιους δείκτες, κάποια κριτήρια που θεσπίζουμε για να δούμε εάν πετυχαίνουμε τους στόχους που έχουμε θέση με την πολιτική μας. Και όσον αφορά τη λογοδοσία, κατόπιν να προσπαθούμε να επισημάνουμε τα δύνατα σημεία του συστήματος. Και έτσι σε όλα τα μέτωπα προσπαθούμε να δούμε πώς θα σημειώσουμε κάποια πρόοδο που χρειάζεται για τόσο πολύ. Ελπίζω σας κάλυψα. Ναι, ναι, λέει η βουλευτής. Τώρα όσον αφορά το θέμα της παιδείας και εκπαίδευσης που έθεσαν πολλοί βουλευτές. Γενικώ δεν είναι αρμοδιότητά μας η παιδεία και η εκπαίδευση. Όπως και για κάποια άλλα που αναφέρατε, όπως κάποια θέματα υγείας και υγιεινής. Απλώς εμείς ε, κάνουμε ό,τι μπορούμε στα πλαίσια της ενωσιακής αρμοδιότητας. και πάρα πολλά είναι θέματα εθνικής αρμοδιότητας. Οπότε, συχνά όταν συζητούμε τέτοια θέματα είναι όταν αυτά τα ζητήματα έχουν να κάνουν με διδύσμες διακρίσεις, με μειονότητες ή με τα δικαιώματα των ανηλίκων. Οπότε δεν έχουμε μια γενικότερη άποψη, έποψη τέλος πάντων του πώς έχουν τα πράγματα στην παιδεία. Πάντως για τους ε, Ρωμά, τους ε, ε, αναπήρους, τους ΛΟΑΔ, για εθνικές μειονότητες, ήταν, είπαμε, θέμα προτεραιότητας η παιδεία. Και έγινε και αυτή η μεγάλη έρευνα για το πώς θα πάει το εκπαιδευτικό σύστημα με αυτές τις κοινωνικές ομάδες. Και εδώ είναι η αδυναμία του τι θα κάνουμε με αυτά τα προβλήματα σε επίπεδο Πολλές φορές βλέπουμε τα πράγματα από πλευράς ε, της μειονότητας και έρχεται κάποιος από την ε, πλειοψηφία από το ΣΥΠΗΝ και λέει μα γιατί και, και εγώ δεν θα με καλύψετε. Το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα μας θα προσπαθήσει να δει πώς μπορούμε να καλύψουμε το σύνολο της κοινωνίας. Παρακάτω τώρα για την ε, ελεύθερη διακίνηση και κάποια θέματα κάποιων στοιχείων όσον αφορά το κοινωνικό dumping που αναφέρθηκε. πολλά θέματα αγοράς εργασίας δεν είναι αρμοδιότητες δικής μας. Είναι όμως όταν έχουμε κάποιες ακραίες μορφές εκμετάλλευσης. Τότε ασχολούμεθα με το πρόβλημα. Πάντως, ό,τι μας απασχολεί τελικά το χρησιμοποιούμε για το πρόβλημα του κοινωνικού ντάμπινγκ. Πώς θα χτενίσουμε την ε, έκθεση, θα δούμε τι γίνεται όσον αφορά τους επιθεωρητές της αγοράς απασχόλησης και θα το κείμενο θα το βελτιώσουμε. Να δούμε επομένω πώς ε, αυτοί οι επιθεωρητές κάνουν τη δουλειά τους, πώς μπορούν να την κάνουν καλύτερα, τι εντολή έχουν, τι έχει διαπιστωθεί. Πάντα βέβαια για τις περιπτώσεις ακραίας εκμετάλλευσης, αλλά βέβαια όλα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και γενικότερα. Τώρα όσον αφορά την παιδεία, είπαμε τα βασικά του προβλήματος. Ούτε εκεί έχουμε τόση πολλή αρμοδιότητα. Τώρα για αυτές 180.000 αυτών των ιονί σκλάβων ε, και τι γίνεται με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας αυτό είναι βεβαίως μια χονδροειδής, μια προσεγγιστική ε, ε, πληροφορία. Δεν έχουμε ακριβείς αστικές. Ίσως, ε, να πούμε και 800.000 με 300-400.000 τελικά. Να είμαστε πιο ρεαλιστές, να μην φουσκώνουμε τα νούμερα. Πάντως, μιλούμε για πολλούς. Πολλούς που ζουν σε συνθήκες σχεδόν σκλαβιάς, δουλειά στην Ευρώπη. Το 2009 ξεκινήσαμε σε συνεργασία με την Europol για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ήμασταν πάρα πολύ απογοητευμένοι γιατί γίνονται πάρα πολύ λίγα σε εθνικό επίπεδο διότι οι διοικητικέ αρχέ, τα κράτη-μέλη όπω και οι επιθεωρητέ εργασία δεν νοιαζόντουσαν για το φαινόμενο. Και από τότε που ξεκινήσαμε έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμο το πρόβλημα, αλλά ακόμα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μα. Στα πολιτικά συστήματα βέβαια τώρα στην Ευρώπη αναγνωρίζονται ότι υπάρχει ένα τέτοιο φαινόμενο. Αλλά ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Τώρα αν αυξήθηκε ή όχι το φαινόμενο ε, δεν μπορούμε να το πούμε και δεν μπορούμε να συγκρίνουμε προηγούμενα αριθμητικά στοιχεία. Έχουμε μόνο τα καινούργια. Κύριε Σιλικιώτη, για αυτό το οποίο ρωτήσατε. Και για τις αιτίε για το ιστορικό πλαίσιο του, του, φαινομένου βάσει της κρίσης και των μέτρων λιτότητας. Τι να σας πω, δεν είναι δουλειά μου να τα σχολιάσω αυτά, αλλά άπαξ και εμείς στην ε, ε, ετήσια έκθεσή μας τα τονίσαμε. Και όπως έλεγα στο τέλος της ομιλίας μου, διαπιστώσαμε κάποια πράγματα. ότι ο οικονομολόγος που ασχολείται με αυτά θα πρέπει να έχει και έναν νομικό ειδικό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Για κάθε βήμα της Τρόικας θα έπρεπε να μελετάτε ο κοινωνικός ε, αντίκτυπος. Τι αντίκτυπο έχουν οι οικονομικές πολιτικές που συζητούνται. Οπότε εξετάζοντα το, αυτό θα μπορούσα να το πω έτσι επιφανειακά, γιατί ούτε τέτοια εντολή έχουμε, ούτε είμαι οικονομολόγος. Αλλά όντω κάποια από τα αρνητικά αποτελέσματα πάνω στον άνθρωπο θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί εάν είχαμε ε, κάποιους να σκέφτονται και τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν σχεδίαζαν τα Μήτρα λιτότητας. Η κυρία, η κυρία Λόπες από την Ισπανία. Ναι, δεν μπορώ να δω καλά τα γράμματα που αναφέρουν το όνομά σας στο κοινοβούλιο, ποτέ δεν τα καταφέρνω. Το θέμα των δύο διαφορετικών φύλων ολώνει και περισσότερο το με υπόψη. Γι' αυτό και στην Ισπανία και σε Εμένα όσον αφορά τη δουλειά μα για την βία κατά των γυναικών. Επομένως και εμείς αυτό θέλουμε να ενταχθεί στις πολιτικές ...στο θέμα ε, των ανισοτήτων. Έχουμε και την υπηρεσία του Βίλνιους που ασχολείται με την ε, ισότητα ή ανισότητες των δύο φύλων. Για τους Ρωμά, Είπαμε τι γίνεται για τους αναπήρους όπως το αναφέρατε κι εσείς. Έχουμε τη βία κατά των ε, αναπήρων, αυτού του είδους τα εγκλήματα μίσους που έχουν στόχο τους αναπήρους και επομένως ε, θα δούμε τι γίνεται και με τους ανηλίκους στο μέλλον ως προς αυτό. κύριος Φουντούλης, σας αναφέραμε ήδη το θέμα της ακραίας ε, εκμετάλλευσης. Και άρα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται σε περίπτωση που οι εργοδότες δεν συμμορφώνονται με τον νόμο. Τότε έχουμε περιπτώσεις ακραίας εκμετάλλευσης. Κύριος Κρασνακόφσκι για τους Ρωμά. Αναφέρεται την πρόσβαση ε, για τις περιπτώσεις υγείας, του, τον εκλογικό νόμο, τι γίνεται στη Γερμανία, ναι. Αλλά, ναι, αυτό είναι από την οπτική γωνία της μειονότητας. Εκεί έχουμε εντολή να εργαζόμαστε. Αλλά όπως είπαμε έχουμε και μια έρευνα για το σύνολο της κοινωνίας, το, η οποία αυτή η έρευνα θα ολοκληρωθεί σύντομα κέντρο για τους αναπήρους στην ε, Γαλλία όσον με την απασχόληση εταιρείε, δεν έχουμε στοιχεία. Ε, δεν ξέρουμε τι γίνεται σε άλλες χώρες. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβληματίζεται όλο ενώ αφορά την εταιρική ευθύνη. Τι κάνουν οι εταιρείε για τα προβλήματα των αναπήρων και άλλα. Θα πρέπει να δώσουν περισσότερη προτεραιότητα οι εταιρείε σε αυτά τα προβλήματα. Εδώ και περίπου 20 χρόνια συζητάμε την ε, εταιρική ευθύνη όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αρκετά το συζητήσαμε, ε, ήρθε η ώρα τα λόγια να γίνουν έργα. Οπότε και γι' αυτό και παρακολουθούμε το πώς πάνε τα πράγματα. Ξέρουμε τι δεν πρέπει να γίνει, πώς θα πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος πιο ζωντανός, Και ύστερα. Τελευταία ερώτηση. Του κυρίου Μάρτιν για τους Ρωμά και το κατά πόσον ε, θέλουν να ενταχθούν, θέλουν να αφομοιωθούν. Καταρχάς, ε, να σας πω ότι οι Ρωμά που συναντώ εγώ και ήμουν σε ένα κρατός μέλος την προηγούμενη εβδομάδα μάλιστα, σε μια συνάντηση με ε, Ρωμά, με το Δήμαρχο, με την πλειοψηφία των πολιτών σε ένα μικρό χωριό, το σαφές μήνυμα είναι ότι θέλουμε να ξεφύγουμε από τη φτώχεια. Θέλουμε να είμαστε τμήματα της κοινωνίας. Άρα είτε το πείτε συμπερίληψη, αφομοίωση, συμπερίληψη ίσως να είναι πιο σωστός όρος, γιατί είναι το πιο ευρύ και ίσως ε, να επιτρέπει και τη διαφοροποίηση. Αυτό που επίσης παρατηρώ όταν επισκέπτομαι χωριά, και άλλους ε, χώρους, αλλά μέρη όπου υπάρχει πληθυσμός Ρωμά είναι ότι η εκπαίδευση και το ποσοστό εκπαίδευσης αυξάνεται. Αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτοί που είναι 20 χρονών σήμερα είναι πολύ καλύτερα εκπαιδευμένοι, έχουν πολύ καλύτερη εκπαίδευση από ό,τι οι γονείς τους. Και πάλι δεν είναι καλό το ποσοστό εκπαίδευσή του. αλλά κινούμαστε προς σωστή κατεύθυνση. Αυτό το επιβεβαιώνουν και τα στατιστικά στοιχεία. Αλλά και οι επισκέψεις μας ε, στις κοινότητε αυτές, στις κοινωνίε αυτές. Ευχαριστώ πολύ, λέει. Και τώρα σας ευχαριστώ κι εγώ, λέει η Πρόεδρος, για τι απαντήσεις αυτές. Σας ευχαριστώ που συμμετείχατε στη διαδικασία αυτή. Uh, uh, και τώρα να περάσουμε στο 5 της ημερησίας διάταξης, το οποίο και συνδέεται αμέσως με αυτά που συζητάμε εδώ για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της της εργασίας. Να δώσω το λόγο παρά αυτά στον κύριο Πυρίνσκι που είναι ο εισηγητής μας από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, το θέμα της αντιμετώπισης της αντίλητης εργασίας συζητείται εδώ και πολλά χρόνια ήδη. Όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το συζητούν και θα ήθελα να πω ευθύς εξ αρχής, Πρόεδρε, ότι έχει έρθει καιρός πια να αναλυθεί δράση. Δράση προκειμένου να αλλάξει η κατάσταση σε ό,τι αφορά την αντίληπτη εργασία, γιατί δεν βελτιώνονται τα πράγματα. Επιδεινώνονται μάλιστα. Πρόκειται για ένα τεράστιο και πολυσύνθετο πρόβλημα. Όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, φαίνεται ότι το θέμα αυτό της αντίληψης εργασίας επηρεάζει με δεσμενή τρόπο την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Άρα θεωρώ ότι έχει φτάσει πραγματικά το πλήρωμα του χρόνου στοχευμένα να καταπολεμήσουμε με δράσεις, με ενέργειες τα συμπτώματα και τις ρίζες, τη γενεσιουργό αιτία του προβλήματος αυτού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ξέρουν οι συνάδελφοι, έχει καταθέσει μια πρωτοβουλία για να τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αθλητικής εργασίας τον Απρίλιο του φετινού έτους. Και το Συμβούλιο συμφώνησε στα μέσα Οκτωβρίου. Τώρα λοιπόν είναι δικό μας καθήκον, δική μας πρόκληση να καθορίσουμε ποια θα είναι η τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να περάσουμε στη φάση διαβούλευσης και να αποφασιστεί, ελπίζουμε, η πλατφόρμα αυτή. Ευθύ εξ αρχή, Πρόεδρε, θα ήθελα να επισημάνω το εξή στου συναδέλφου. Στόχο, θεωρώ, θα πρέπει. Και αυτό θα πρέπει να καθορίζει όλες μας τις δράσεις σε ό,τι αφορά το ψήφισμα είναι να κάνουμε διαφορά. Τη διαφορά στην σελίδα 20, τροπολογία 45, αυτό αναφέρεται σε μια τροπολογία που προτείνω να εγκρίνουμε ότι ο απότερος σκοπός θα πρέπει να είναι η πλατφόρμα αυτή να παράσχει προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα κράτη-μέλη και στα συνδικάτα προκειμένου με συνεργασία να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το θέμα της αδρέτης εργασίας. Και πάλι λοιπόν σε ό,τι αφορά την προηγούμενη παρουσίαση θα προσέξετε όλοι φαντάζομαι το γεγονός ότι το πρόβλημα που αναφέρθηκε σε ό,τι αφορά τους επιθεωρητές εργασίας και τη μειούμενη αποδοτικότητά τους. Πολύ ανησυχητικό το φαινόμενο αυτό, καθότι ξέρουμε ότι η εμπειρία των ε, υψηλόβαθμων ε, επιθεωρητών συνέβαλε σημαντικά στις προσπάθειες των κρατών μελών προκειμένου να τηρείται καλύτερα το εργατικό δίκαιο συμπεριλαμβανομένου και του θέματος της αδελφής εργασίας. Και πάλι να υπογραμμίσω μια επιπρόσθετη διάσταση. Πολύ απαραίτητη θεωρώ, προκειμένου η πλατφόρμα αυτή να καταστεί πιο αποτελεσματική και αποδοτική η έννοια της ε, νομιμοποίησης ε, ε, της μαύρης εργασίας. Αυτό λοιπόν θα νομιμοποιήσει, θα φέρει στην κανονική αγορά εργασίας κάποιες ε, θέσεις απασχόλησης που είναι στη σκιώδη οικονομία σήμερα. Και να είμαι σαφής σε ό,τι αφορά ένα στοιχείο της νομιμοποίησης. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί, να ερμηνευθεί ως δικαιολογία για διαφόρων ειδών επισφαλούς απασχόλησης. Μερικής απασχόλησης ε, σε επισφαλείς όρους, με χαμηλό μισθό και μάλιστα με τέτοιο τρόπο ώστε να νομιμοποιηθεί τελικά η εκμετάλλευση σε καμία περίπτωση δεν, αποσκοπώ, δεν έχω αυτό σκοπό όταν προτείνω το στοιχείο αυτό στην πλατφόρμα. Ανακύπτει λοιπόν πάρα αυτό το ερώτημα του πώς θα λειτουργήσει αυτή η πλατφόρμα, τι είδου δραστηριότητες, τι είδου καθήκοντα θα πρέπει να εμπεριέχει. Εδώ υπάρχει κάποιος δισταγμός, κάποια διστακτικότητα από τα κρατημέλη, απροθυμία σε ό,τι αφορά λήψη αποφάσεων για υποχρεωτικά μέτρα λίγο πολύ. που θα εξαναγκάσουν τα κρατημέλη να κινηθούν προς μια κατεύθυνση την οποία δεν επιθυμούν. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να σας καλέσω και όλους αυτούς όσοι ασχολούνται με το θέμα αυτό να το εξετάσετε αυτό ως μια κοινή προσπάθεια. Μια κοινή προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων των κυβερνήσεων, γιατί αυτό αφορά και τα θέματα κοινωνικών επιδομάτων, φορολογικής, ε, φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής, των ε, εργατικών κινημάτων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμμετάσχουν σε μια προσπάθεια κατάργησης του κοινωνικού ντάμπινγκ και του επιχειρηματικού κόσμου που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να απέφχονται τον αφέμητο ανταγωνισμό. Αυτό λοιπόν που έχει ως σκοπό η πλατφόρμα είναι να υπάρχουν έγκυροι εκπρόσωποι από τις κυβερνήσεις, από τους εργοδότες και τους εργαζόμενους, από ευρωπαϊκά σώματα, προκειμένου καταρχάς να υπάρξει μια ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Ύστερα, να, υπάρχουν, να υπάρξουν λύσεις που έχουν αποδειχθεί επιτυχή σε ό,τι αφορά την πρόληψη και την νομοποίηση της αντρεύης εργασίας. Πολλά τέτοια παραδείγματα υπάρχουν, τα οποία και συνάντησα κατά την προετοιμασία της έκθεσης αυτές. Πολύ χρήσιμο θα ήταν να τα γνωρίζουν όλα τα κρατη και όλα τα θεσμικά όργανα, προκειμένου να δουν τι μπορούν να εφαρμόσουν και τι μπορούν να βελτιώσουν. Υπάρχουν διάφορα πρακτικά ζητήματα σε ό,τι αφορά την πλατφόρμα αυτή, πώς θα οργανωθούν οι εργασίες της, πόσο συχνά θα συναντιέται, σε ποιον θα υποβάλει αναφορά. Δεν θέλω να σας κουράσω και να μακρηγορήσω. Το μόνο που θα ήθελα παράλληλα αυτά να επισημάνω είναι ότι έχουμε την αίσθηση ότι το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας θα πρέπει να συμμετάσχουν και να παρακολουθούν τις δραστηριότητες της πλατφόρμας προκειμένου να κινηθεί στην κατεύθυνση την οποία και περιέγραψα. Και κλείνοντας θα ήθελα και πάλι να ξεκινήσω, να τελειώσω από εκεί που ξεκίνησα, από το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, γιατί έχουμε μία τροπολογία αγαπητοί Πρόεδρε, την υπαριθμόν και αναφέρει ότι το έργο της πλατφόρμας θα πρέπει να σέβεται το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και συγκεκριμένα άρθρα συγκεκριμένα 5.15.51 καθώς και τις σχετικές συνθήκες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας. Και υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν θα ήθελα να σας ζητήσω να εξετάσετε την έκταση αυτή. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος, ευχαριστώ με τον κύριο Πυρίνης και να ξεκινήσουμε τώρα με τη Ρεμάνα Τόμψ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Πυρίνσκι για την τόσο σφαιρική έκθεση που έχει συντάξει. Είναι πολλές οι τροπολογίες, 71. Αυτό σημαίνει ότι έχουν γίνει ήδη πολλές σοβαρές προσπάθειες για να βελτιωθεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά την άποψή μου, η πρόταση η ίδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ καλή βάση και επιδιώκει τους ίδιους ε, στόχους που και εμείς επιθυμούμε να φτάσουμε. Μπορεί κάποιες φορές οι απόψεις μας για τις λύσεις ε, που προκρίνουμε να διαφέρουν, αλλά μπορούμε να βρούμε συμβαστικές λύσεις και τελικά έχουμε ένα κοινό στόχο. Να αποτρέψουμε, να μειώσουμε και να εξαλείψουμε την αδήλωτη εργασία σε κάθε κράτο μέλος. Αυτή η πλατφόρμα λοιπόν είναι ένα από τα εργαλεία που θα έχουμε στα χέρια μας για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Για να μειώσουμε τα επίπεδα της αδήλωτης εργασίας. Βεβαίως, είναι σημαντικό η πλατφόρμα αυτή να μην γίνει αυτός ο σκοπός. Να λειτουργεί πραγματικά και στην πράξη, σε καθημερινότητα. Είναι σαφές ότι οι τροπολογίες του κυρίου Πυρίνσκι υπό πολλές απόψεις πάνε ακόμη πιο μακριά από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προβλέπουν κάποιες νέες έννοιες όπως την νομιμοποίηση. Αυτά είναι θέματα που θα τα συζητήσουμε ξανά. Και είμαι πεπισμένη ότι παρά τη σκληρή δουλειά που έχουμε μπροστά μας, για ένα τόσο σύντομο κείμενο, τουλάχιστον έχουμε κοινού στόχους. Και επίσης πιστεύω και είμαι πεπισμένη ότι θα πετύχουμε να βρούμε συμβαστικές λύσεις ώστε να μπορέσουμε αυτό το κείμενο να το εφαρμόσουμε και στην πράξη. Δεν θέλουμε να παραμείνει μόνο στα ωραία λόγια, αλλά να υπάρχει επιτυχής συνεργασία. Ευχαριστώ. Πρόεδρο. Ευχαριστούμε ο κύριος Καρατσάμπο από την ομάδα των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας μιλώ εκ μέρου κυρία που είναι η σκιώδη συζητητριά μας. Δεν μπόρεσε να παραστεί. Οπότε επαναλαμβάνω ότι σας λέγω ε, αυτά τα οποία εκείνη πρεσβεύεται και δεν ε, συμφωνούμε πάντοτε και αναγκαστικά. Πάντως τον θέλει να σας πει ότι πρόκειται για κάποια προσθεμένη αξία επειδή παρά το ότι βρισκόμαστε σε κάποια πάρα πολύ δύσκολη φορολογική, δημοσιονομική ε, συγκυρία που περνάνε όλες οι χώρες οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλο της Επιτροπής και εμείς ως Άλντε παρακολουθούμε τις εξελίξεις και η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κάτι που μας βρίσκει συμφώνους και Παρ' όλα αυτά εμείς θα θέλαμε να εμπλουτιστούν οι απόψεις με κάποιο είδους πιο, πιο σφαιρική ε, αντιμετώπιση του προβλήματος. Δηλαδή να ρίξουμε μυθιά και στα δημοσιονομικά για το πώς θα έχουμε καλύτερη νομοπαρασκευαστική ποιότητα, ε, καλύτερη διοίκηση και ε, διοικητική διαχείριση. Ε, συμφωνούμε βέβαια με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ότι πρέπει να εμπλακούν τα κράτη-μέλη και αυτά που δεν έχουν εμπλακεί ακόμα. Θα πρέπει επίσης να εμπλέξουμε εδώ και διάφορους φορείς και κατά νου έχω τώρα την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της χώρας μου. Ακόμα δεν έχουμε τοποθετηθεί όσον αφορά τι γίνεται με τους ελεύθερους επαγγελματίε και τι σχέση έχει, ε, τι σχέση έχει αυτός ο κλάδος με ε, την παραοικονομία. Παναβάνω, μιλώ για σκιώδη συγγήτρια. Από πλευράς της θέλω να σα πω ότι θα πρέπει αυτή η πλατφόρμα να προχωρήσει και να καταστεί με τη διαχείριση του ζητήματος των επιθεωρητών εργασίας, οι οποίοι θα πρέπει να επιβληθούν κατά κάποιο τρόπο στα κρατημέλη, στις πατρίδες τους. Και φυσικά δεν τα λέμε όλα αυτά ενάντια στην αρχή της επικουρικότητας. συμφωνούμε με όλα όσα αναφέρθηκαν ότι πρέπει να γίνουν, αλλά επίσης και θα θέλαμε να μην έχουμε περισσότερο διοικητικό άχθος στις επιχειρήσεις, να μην βάζουμε περισσότερη γραφειοκρατία, τα πράγματα, τη διοίκηση ε, και να μην παρεμποτίζεται το έργο των ΜΜΕ. Σας ευχαριστώ. Από τους συντηρητικούς μεταρρυθμιστές, κύριε Μακιντάερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Πυρίνσκι, τον εισηγητή, για όλη τη δουλειά που έχει κάνει ως τώρα. Και καλωσορίζουμε την δημιουργία μιας τέτοιας πλατφόρμας. Είναι σημαντικό να μπορούμε να ανταλλάξουμε τις βέλτιστες πρακτικές και τις ανάλογες πληροφορίες και να υπάρχει και μια κοινή κατανόηση για το τι είναι αδειλωτή εργασία. Είναι μια άριστη ευκαιρία ώστε τα κράτη-μέλη να ξεκινήσουν ε, ε, εντατική διασυνοριακή συνεργασία και την ε, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα για όλα τα κράτη-μέλη, ιδίως ως προς δύο τομείς της φοροδιαφυγής και του αθέμετου ανταγωνισμού, αλλά και για την προστασία των εργαζομένων και την ασφάλειά τους. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό ζήτημα. Τώρα για την φύση της αδειλωτής εργασίας. Ξέρουμε ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Νομίζω πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε μία ακριβώς, ακριβή λύση για όλους την ίδια. Από τη δική μου εμπειρία, στη δική μου χώρα, αδήλωτη εργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι περίπου 1,7% βάσει των στοιχείων του ΩΣΑ σε άλλα κράτη-μέλη είναι πολύ ψηλότερα τα ποσοστά. Νομίζω λοιπόν, όταν κοιτάζουμε την ε, συμμετοχή, ένα θέμα που το είχαμε ήδη συζητήσει, εάν θέλαμε, αν θέλουμε να υπάρξει υποχρεωτική συμμετοχή και είμαι θετική ως προς αυτή τη λύση, διότι αν θέλουμε αυτό να πετύχει όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δεχτούν την υποχρεωτική συμμετοχή. Εάν το κάνουμε λοιπόν αυτό, το να μην υπάρχει διεξοδικός κατάλογος υποχρεωτικών δράσεων γίνεται ανέφικτο. Ίσως χρειαστεί πρώτα απ' όλα η υποχρεωτική συμμετοχή από τη μία σύστημα και μετά κράτη-μέλη να δικαιολογούνται στις επιμέρους ενέργειες για το τι δεν θέλουν συμμετοχή σε μία συγκεκριμένη ενέργεια. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε δεσμευτική συμμετοχή και μη διεξοδικό κατάλογο. Δεν γίνεται αυτό, να μην ξέρουμε τι θα θέλουν να κάνουν τα κράτη-μέλη που οπωσδήποτε θα συμμετέχουν. Έχουμε επίση και κάποιε ανησυχίε για την ε, εισαγωγή αυτή τη έννοια, τη νομιμοποίηση τη εργασία, regularization στα αγγλικά. Ε, θέλαμε διευκρινήσει ω προ το τι σημαίνει αυτό. Τι ακριβώ δεν εννοεί ο συγητή, αν μπορεί να μα πει. Δηλαδή τι αποκλεί αυτός ο ορισμός, για να καταλάβω έτσι κάτι ακριβώς θέλει να πει. Αν μας πει ότι δεν εννοεί, ίσως θα έπρεπε λίγο να αλλάξουμε τη διατύπωση για να είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που λέτε. Γιατί για μένα διευρύνει πάρα πολύ το ε, πεδίο που θέλουμε να καλύψουμε και αυτό κάπως με ανησυχεί. Και ένα-δυο ακόμη σχόλια. Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Σωστά τα λέτε, ιδίω σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά τι θα γίνει εάν πούμε στα κράτη-μέλη τι πρέπει να κάνουν ω προ τι διαβουλευσει προτού προσέλθουν σε συνεδρίαση και του πούμε ποιον πρέπει να φέρουν μαζί τους. Εδώ λιγάκι θα προσπαθήσουμε να διευθύνουμε υπερβολικά τα πράγματα και αυτό δεν νομίζω ότι θα πετύχει. Και κάτι ακόμη. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προσέξουμε τι προτάσεις κάνουμε για την ανταλλαγή δεδομένων. Υπάρχει ειδικό ε, καθεστώς για κάποιο είδου πληροφορίε, όπως τις φορολογικές. Αυτό θα προκαλέσει έτσι κι αλλιώς δυσκολίε στην ανταλλαγή δεδομένων. Οπότε ας είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς θα χαρακτηρίσουμε τα διάφορα δεδομένα και το τι ακριβώς θα ε, ε, απαιτηθεί. Όπως φαντάζεστε. Νομίζω και εγώ έχουμε πολλές, ε, πολλούς γύρους διαπραγματεύσεων μπροστά μας, όμως ε, είμαι και εγώ θετική στο να βρεθούν συμβαστικές λύσεις και θα κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω. Ευχαριστούμε κυρία Κούνεβα από την ΒΟΕ. Ε, Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχαίρω τον εισηγητή τον κύριο Πίδινσκι για την πολύ καλή έκθεσή του. Είναι πολύ σημαντική η προσέγγιση που υιοθετεί συμφωνώ να πάμε ένα βήμα παραπέρα από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όχι μόνο καταγραφή και πρόληψη του προβλήματος που έχει βατίες οικονομικές και κοινωνικές ρίζες. Να βοηθήσουμε και στην μετατροπή της παράνομης εργασίας σε νόμιμη και καταγεγραμμένη εργασία Χαίρομαι επιπλέον γιατί συμφωνούμε να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των κράτων στην πλατφόρμα. Γιατί αν είμαστε αποφασισμένοι να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο δεν πρέπει να αφήσουμε περιτόρια για κοινωνικό dumping. Βρίσκω πολύ σωστή και την ιδέα χατορισμού ενός από κάθε κράτος που θα συντονίζει τις εθνικές δράσεις για την αντίλωτη εργασία σε συνεργασία πάντα με τους άλλους αρμόδιους φορείς. Ο εκπρόσωπος αυτός όμως δεν είναι απαραίτητο να είναι κυβερνητικός, αλλά πρόσωπο με εμπειρία και αποδοχή. Πολύ σωστή είναι και πρόταση για κοινή προσέγγιση από τα κράτη-μέλη των εταιριών που χρησιμοποίησαν, αντίλο, που χρησιμοποίησαν Και εδώ τα κοινά μέτρα δεν αφήνουν περιθώρια εκμετάλλευσης μιας ευνοϊκότερης νομοθεσίας για τους παραβάτες. Χρήσιμη βλέπω και την πρόταση για καλύτερη εσωτερική οργάνωση της πλατφόρμας με τις θεματικές ομάδες εργασίας. Ωστόσο, Χρειαζόμαστε ένα άλλο ορισμό της αντιδότης εργασίας. Δουλεύουμε με έναν ορισμό το 1998 και αναρωτιέμαι αν αυτό είναι λογικό. Η προτεραιότητα της πλατφόρμας πρέπει να καλύψει σε έναν ορισμό που περιγράφει τα σύγχρονα φαινόμενα και τα πολλά πρόσωπα που παίρνουν σήμερα η αντιλωτή εργασία. Τι εννοώ. Λόγω των ιδιωτικών μέτρων που επιβάλλουν, διοικητικών μέτρων που επιβάλλουν κάποια κράτη-μέλη σε εργοδότες και επιχειρήσεις που απασχολούν αντίλωτου εργαζόμενους, αντιμετωπίζουμε φαινόμενα της μερικής αντίλωτη εργασίας Δηλαδή κάποιοι εργοδότες αναγκάζονται μεν να δηλώσουν τους εργαζόμενους τους, αλλά όταν το κάνουν αποκρύπτουν όλες τις ώρες εργασίας και δεν αποτυπώνουν πλήρως το πραγματικό καθεστώς απασχόλησης και ασφάλισης τους. Αυτό όχι μόνο δεν ονίζει τα προβλήματα που θέλουμε να αποφύγουμε, αλλά έχει και σαν αποτέλεσμα την βελτίωση των εθνικών δικτών με τρόπο πλασματικό. Έτσι, κυβερνήσεις όπως η ελληνική επιχαίρει για παράδειγμα για μείωση της ασφαλιστικής εργασίας όταν είναι προφανές ότι απλώς οι εργοδότες και πάλι δηλώνουν τη μισή αλήθεια. Δημιουργείται δηλαδή ένας φαύλος κύκλος που επιθύνει το φαινόμενο χωρίς ωστόσο αυτό να είναι εμφανές. Θα υποβάλω σχετική τροπολογία και θα παρακαλούσα τον εισηγητή να δει αυτό το θέμα με μεγάλη προσοχή. Επιπλέον, ως εισηγήτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Ισότητας και Δικαιωμάτων των Γυναικών, έχω προτείνει τροπολογίες που αφορούν την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δώσουμε στις γυναίκες που είναι τα συχνότερα θύματα της εργασίας όσον αφορά τη δουλεία, δουλειά στο σπίτι και σε μεγαλύτερους ανθρώπους. Ελπίζω μια καλή συνεργασία και σας ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. ειδάκια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, Νομίζω ότι πολλά σημαντικά στοιχεία ήδη αναφέρθηκαν στη συζήτηση. Να ευχαριστήσω καταρχάς τον κύριο Πυρίνσκι για το γεγονός ότι ως κοιόδης είχαμε ήδη την ευκαιρία να έχουμε μια συνάντηση και να συζητήσουμε τις ιδέες μας. Τρία σημεία θα ήθελα να προσθέσω που πιστεύω ότι χρειάζεται διευκρίνηση ή και προσθήκη στην πρόταση. Πρώτον, πιστεύω ότι αν υπάρξει πλατφόρμα και αν υποτίθεται ότι ο σκοπός μας είναι να αποτελεί ένα σημείο συντονισμένης δράσης ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλους τους εμπειρογνώμονες και τους εμπλεκόμενους φορείς και σε ό,τι αφορά την αντίλατη εργασία. Γιατί ιδάλλως υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει μια παράλληλη εργασία με άλλες ομάδες εμπειρογνωμόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προκειμένου λοιπόν να μην γίνει αυτό, να συμπεριληφθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και όλοι οι εμπειρογνώμονες. Πολύ κρίσιμο σημείο. Δεύτερο στοιχείο και στις προηγούμενες συζητήσεις αναφέρθηκε αυτό σε διάφορες περιπτώσεις, σε διάφορες περιστάσεις, ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει μόνο ανταλλαγή απόψεων και τελικά να μην γίνεται τίποτα. Όχι, χρειάζεται σαφείς στόχους, σαφή καθήκοντα η πλατφόρμα. Και νομίζω ότι εδώ χρειάζεται κάποια διευκρίνηση για το τι συμπεριλαμβάνεται ήδη σήμερα στην πλατφόρμα συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων δράσεων σε επίπεδο κράτους μέλος, όχι δηλαδή μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να διευκρινιστεί ότι σε κάποια πράγματα και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συντονιστούν, να συντονίζουν τις δράσεις τους. Και για να το πατήχουμε αυτό θα πρέπει τα κρατημέλη να δείχνουν την ανάλογη προθυμία. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. Sven Schulze. Ευχαριστώ κύριε Σβέν Σούλτσε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πυρίνσκι για τη δουλειά που έκανε. Είναι πολύ καλό το σχέδιο έκθεσης ήδη. Και εγώ να πω ότι ήδη Ακούσαμε από τους προλαλήσαντες πολλά σημαντικά σωστά στοιχεία και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι από πλευρά μου χρειαζόμαστε δεσμευτική συμμετοχή των κρατών μελών γιατί νομίζω ότι η καταπολέμηση της αντίληψης εργασίας θα φέρει περισσότερη δικαιοσύνη σε κάθε κράτος μέλος. Αυτούς που σηκώνονται κάθε πρωί πάνε στη δουλειά τους και πληρώνουν τους φόρους τους όπως προβλέπεται στο κάθε κράτος μέλος. αλλά πιστεύω ότι στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις για το τι, αποτελεί αδήλωτη εργασία. Υπάρχουν και διάφορες διαφορετικές δομές καταπολέμησης. Δεν υπάρχει ένας ε, οριστικός ορισμός της αδήλωτης εργασίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι η πλατφόρμα αυτή θα έχει πιο πολύ ενημερωτικό χαρακτήρα για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Και ύστερα θα πρέπει οι αρμοδιότητες να παραμένουν σε επίπεδο κράτους μέλους. Επίσης, θεωρώ ότι είναι πολύ καλό σε ό,τι αφορά τις ιδέες που περιλαμβάνονται στο έγγραφο του Συμβουλίου, στο 11α, 11β, να τις τονίσουμε και να επανέλθω στο άρθρο 11 της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί θεωρώ ότι αυτό το άρθρο που αφορά θέματα παρακολούθησης και ελέγχου δεν πηγαίνει αρκετά μακριά, μέχρι εκεί που πρέπει. Θα πρέπει να οριστεί καλύτερα. Ίσως να υποβάλλω σχετική τροπολογία. Κάτι άλλο που είναι για μένα σημαντικό και επίσης αναφέρθηκε από τους συναδέλφους ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η πλατφόρμα αυτή θα περιλαμβάνει εκπροσώπους υψηλό βαθμούς από τα κράτη-μέλη προκειμένου να μην αποτελέσει μία πλατφόρμα, άλλη μία πλατφόρμα από τις πολλές. Θέλουμε λοιπόν καλά εκπαιδευμένους εμπειρογνώμονες στην πλατφόρμα αυτή. Μαρτά, ευχαριστώ. Παρόλο που δεν συμμετείχαμε σε όλη αυτήν την δουλειά, την ετοιμασία της ε, ευχαριστούμε τον κύριο Πυρίσκη για όσα μας προτείνει. Βεβαίως, πρέπει να προβλέψουμε κάτι για να καταπολεμήσουμε την αδύλατη εργασία. Την όμως, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Η πίεση της ε, δημοσιονομικής πολιτικής λιτότητας ουσιαστικά πιέζει και τη μία πλευρά του εργοδότη και του εργαζομένου, οι οποίοι προσπαθούν να επιβιώσουν, να συνεχίσουν απλώς να υπάρχουν. Οι επιχειρήσεις τι δυνατότητες έχουν εξαιτία της δημοσιονομικής ασπίεσης και της φορολογίας της λιτότητας, να κηρύξουν πτώχευση και να εξαφανιστούν ή να μετατοπιστούν εις βάρος των ε, εργαζομένων των κρατών μελών ή να χρησιμοποιήσουν σε απόσπαση εργαζομένους, αποσπασμένους δηλαδή, Γάλλοι να πάρουν εργαζομένους που μπορούν να τους πληρώσουν 4 ευρώ αντί για 15 ως 20 με όλη την εξοικονόμηση των ε, κοινωνικών επιδομάτων. Οπότε στα δημόσια έργα με ανεξάρτητους εργαζομένους ή τα νοικοκυριά μπορούν να καλέσουν να φέρουν ε, αδήλωτους εργαζομένους. Τώρα για τον αδήλωτο τον εργαζόμενο το είναι ίδιο ή μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κοινωνικά επιδόματα ως τώρα, τα οποία όμως διαρκώς μειώνονται επειδή η πολιτική λιτότητα σε εξακολουθεί, οπότε δεν μένουν και πολλά, ή έχει το δικαίωμα παρόλα αυτά να αναζητήσει τα μέσα για να γεμίσει το ψυγείο του και να έχει κάτι να φάει ο ίδιος και τα παιδιά του. Ή να πάει στα συσίτια του τοχοκομείου. Οπότε οι πολιτικές λιτότητας και υπερβολικής φρολόγησης που εσείς επιβάλλετε πιέζουν και τα δύο άκρα του συστήματος και την πλευρά των εργοδοτών και των εργαζομένων οι οποίοι ουσιαστικά καταλήγουν στην αδήλωτη εργασία. Μπορείτε να προβλέψετε ό,τι θέλετε ως μέτρο αλλά όταν μιλάμε για επιχειρήσεις ή για εργαζομένους και όταν απλώς προσπαθούν να επιβιώσουν δεν θα υπάρξει άλλος τρόπος. Απλώς θα έχουν μια ε, τέτοια συμπεριφορά μέχρι να υπάρξει μια πολιτική για την ανάκαμψη Τη της οικονομίας και να εξαλείψουμε τη λιτότητα και την ε, υπερφορολόγηση. Thank you, Mr. Ευχαριστούμε κύριο Μπενιφέη. Thank you, Chair. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αρχίζω λέγοντα κάτι για τον κύριο Πυρίνσκι. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά για το σχέδιο της ε, έκθεσης πάρα πολύ στέρεη βάση και αφετηρία για τη συζήτηση. Το είπαν και άλλοι συνάδελφοι. Συμφωνώ με τα περισσότερα που είπε ο εισηγητής μας και με τη γενικότερη του προσέγγιση για το θέμα μας. Επίσης συμφωνώ 100% με το ότι θα πρέπει να εστιάσουμε καλύτερα την προσοχή μας για το έγγραφο όσον αφορά το ζήτημα ε, της καταγραφής των ε, εργαζομένων, των αδήλωτων και άρα θα πρέπει να βελτιωθούν τα πράγματα όσον αφορά την απασχόληση των Ευρωπαίων θα πρέπει να υπάρχει ευκαιρία για αξιοπρεπή δουλειά. Και να έχουμε θέσει απασχόληση, να βγούμε από την κρίση, οπότε και η πλατφόρμα θα πρέπει όλα αυτά να τα έχει προτεραιότητες και να τα φροντίζει, οπότε γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα παραμείνει η πλατφόρμα αυτή αποτελεσματική μια που είναι μια ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Αυτό σημαίνει ότι όλα αυτά θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά, να είναι απλά, λειτουργικά, φιλόδοξα, ε, ιδίω όταν έρθει η ώρα εξαγωγής συμπερασμάτων. Να έχουμε διαφάνεια, να μην αφήνουμε απ' έξω τίποτα, να έχουμε διάδραση, εμπλοκή των κοινωνικών παραγόντων, των θεσμικών οργάνων, των φορέων. Πολύ σημαντικό η κοινωνικοί εταίροι να κάτσουν στο τραπέζι των συζητήσεων και να βρεθεί και ένας, ε, ένας λόγος για το δίκτυο των δημοσίων κρατικών υπηρεσιών, να έχουμε συνέργεια επομένω, να έχουμε συνεργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο με όλα τα δίκτυα, τα υπάρχοντα. Ακριβώς αυτό θέλουμε να πούμε με αυτή τη φράση της συνεργασίας και να πρόκειται για συνεργασία υποχρεωτική, ούτω ως πλατφόρμα να μην χάσει τον προσνοτισμό της. Και έτσι να πετύχουμε τους κοινούς στόχους. Ιδίως όταν έχουμε κάποιο είδους λύσεις για τον ανταγωνισμό, για το κοινικό dumping, για την λαθρομετανάστευση. Πολύ σημαντικά για πιο συντηρητικούς συναδέλφους. Α, είναι πολύ σημαντικά θέματα αυτά και για τους συναδέλφους από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αν και αυτοί συνεργαστούν θα πάει καλά η πλατφόρμα. Όπως όμως το είπε ο κύριος Πυρίνσκι πριν από λίγο. βασικός στόχος είναι να βοηθήσουμε να αντιμετωπιστεί ο αθέμητος ανταγωνισμός από την αντίλωτη εργασία. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο η πλατφόρμα. Να βρεθούν τρόποι να γνωμοδοτεί η πλατφόρμα, να συντάσσει εκθέσεις, τα θεσμικά όργανα να τις ε, ε, μελετούν. Ανάλυση, πρακτικές προτάσεις για την καταπολέμηση της αθλητικής εργασίας. Να καλύψουν τους κοινωνικούς δείκτες στο εξάμεινο το ευρωπαϊκό. Έτσι η πλατφόρμα θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Thank you very much. And now it's Mr. Lenners. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, allereerst... Lenners. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ ικανοποιημένοι αισθανόμαστε από αυτή την πρόταση. Νομίζω ότι είχαμε τη μελέτη τη βιωσιμότητας πριν από τρία-τέσσερα χρόνια, άρα ήταν καιρός να δούμε για την έκθεση του κυρίου Πυρίνσκη. Είπαμε ότι δεν είναι τόσο φιλόδοξη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπήρξε κάποια απογοήτευση και έχω να σας πω ότι μπορούμε να είμαστε ακόμα πιο φιλόδοξοι. Μία από τις λειτουργίες της πλατφόρμας είναι να δούμε το πώς να έχουμε καλύτερη ροή δεδομένων, σημαντικό πρόβλημα, το αντιμετωπίσουμε, την αδίλωτη εργασία, τι γίνεται με, τους, ε, με τα ελευθερία επαγγέλματα, τους εξαρτήτους εργαζομένους, τους αυτοαπασχολούμενους, άρα θα πρέπει να δούμε όρημα το πράγμα. Σε, σε ένα ψήφισμα Είχαμε ζητήσει να υπάρξει μια πλατφόρμα για να καταπολεμηθεί η παραμή εργασία, δίωτη εργασία κλπ. Πολύ σημαντικά είναι αυτά, οπότε σε αυτή τη δέσμη προτάσεων, αυτό το οποίο δεν ρυθμίζεται είναι ο συμβουλευτικός ρόλος, η συμβουλευτική αρμοδιότητα της πλατφόρμας. Είπαμε ότι μπορούν να υποβάλουν συστάσεις, αλλά θα πρέπει κάπως να βελτιώσουμε τη διατύπωση η πλατφόρμα σύντομα να μπει σε λειτουργία. Έχουμε καλύτερη λειτουργία και καλύτερη πρικοδότηση υπηρετές εργασίας. Αυτό πρέπει να το ρυθμίσουν τα κράτη-μέλη. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι. και όπως είπε ο συνάδελφος θα πρέπει να μείνουν νεκρό γράμμα. Το Κοινοβούλιο να παρακολουθεί την πορεία. Μην το παρακάνουμε όσον αφορά τη θεσμική ρύθμιση αυτού του φορέα. Έτσι θα γίνει δυσκίνητος. Αντιθέτως, προσέξουμε πώς θα υπάρξει μια ευέλικτη προσέγγιση πώς θα έχουμε πραγματικά προστιθέμενη αξία. Αν έχουμε χρόνο, λέει Πρόεδρος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να υποβάλει κάποιες προτάσεις για να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ ιδιαίτερος τον συγκητή για την αφοσίωση με την οποία δούλεψες αυτό το θέμα και για την τόσο καλή ε, αντίληψη της κατεπίγουσας κατάστασης και της ανάγκης δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να υπάρξει συνεργασία και να ε, παράγουμε προστιθέμενη αξία σε σχέση με όσα ως τώρα ισχύουν. Ευχαριστώ λοιπόν τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ε, επιδίωξή της να δημιουργηθεί αυτή η πλατφόρμα. Δεδομένων βεβαίως των ε, αναντήρητων αποκλήσεων μεταξύ των κρατών μελών. Θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική συμμετοχή για όλα τα κρατημέλη σε αυτή την πλατφόρμα. Τρεις παρατηρήσεις θα κάνω. Μια πρώτη για τους στόχους. Επανέρχομαι στους κεντρικούς στόχους της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι να ε, ευνοήσει την συνεργασία των κρατών μελών και των αντιφερομένων φορέων για να υλοποιήσουν αποτελεσματικότερα τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους και ως προς την πρόληψη αλλά και την ε, επιβολή κυρώσεων για την αδίλωτη εργασία. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τεχνικά και όλους τους αρμόδιους φορείς των κρατών μελών που καταπολεμούν την αδήλωτη εργασία. Γι' αυτό, όπως το πρότεινε μία βουλευτής, το θέμα διατύπωσης του στόχου της καταγραφής ή νομιμοποίησης των αδήλωτων εργαζομένων θα πρέπει να ε, βελτιωθεί ίσως από την πλευρά του, του λεξιλογίου. Ένας από τους στόχους της πλατφόρμας είναι βεβαίως να στηρίξει την επίσημη αγορά εργασια την νόμιμη αγορά εργασια Το θέμα της νομιμοποίησης λοιπόν ή της καταγραφή τη αδειλότητας εργασίας είναι βεβαίω θεμητό και πολλά κράτη-μέλη έχουν τέτοιου είδους εμπειρίες με νομιμοποίηση ή αμνηστία τρόπον τεινά και οι οποίες θα περιληφθούν σχετικές πληροφορίες στην πλατφόρμα. Απαντούν σε συγκεκριμένε ανάγκε όμω των κρατών μελών και ιδίω για συγκεκριμένου τομεί. Δεν είμαι πάντω βεβαία ότι είναι λύση για όλου του επαγγελματικού κλάδου. Θα πρέπει λοιπόν κάπως να το σκεφτούμε περισσότερο. Ε, έπειτα είδαμε ο εισηγητής να θέλει ενίσχυση του ρόλου των επιθεωρητών εργασία. Είναι όντω μια σημαντική πτυχή μεταξύ των εργαλείων που διαθέτουν τα κρατημέλη για να εντοπίσουν και να προλάβουν την αδήλωτη εργασία. Να θυμίσω όμως ότι ο στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι όχι μόνο να δουλέψουν περισσότερο οι επιθεωρητές εργασίας των κατών μελών, διότι του αυτού του είδους οι επιθεωρήσεις Δεν γίνονται ποτέ από του αρμόδιου για την αδήλωτη εργασία, αλλά θέλουμε να υπάρξει επαγρύπνηση από τα διάφορα σωματεία για τους διάφορους επαγγελματικούς κλάδους. Δηλαδή να υπάρξει μια σφαιρική μορφή συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές και για την φορολογία, τη μετανάστευση, την υγεία στο χώρο εργασίας και την ασφάλεια όλα αυτά να συνδυαστούν για να μην δίνεται η εντύπωση ότι μόνον οι επιθεωρητές εργασίας θα πρέπει να αναλάβουν αρμοδιότητες και ευθύνες για τη λειτουργία της πλατφόρμας. Και τρίτη παρατήρηση, το θέμα της διαχείρισης, της διακυβέρνησης. Υπάρχουν πολλοί ε, που εμπλέκονται εδώ και πολλοί τους οποίους αφορούν οι τροπολογίες του εισηγητού να θυμίσω, όπως το είπαν και κάποιοι από τους παρεμβαίνοντες, μας ενδιαφέρει να παραχθεί προς τη θεμένη αξία, αλλά να είναι και αποτελεσματική η πλατφόρμα στη λειτουργία της. Και επίσης να υπάρχει μια γενική συνοχή στις ε, δράσεις αυτής της πλατφόρμας. Ε, βεβαίως, δεν θα σας ε, διέφυγε ότι βάσει των τροπολογιών του εισηγητή θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική συμμετοχή στην πλατφόρμα. Να τονίσω ότι πιστεύω αυτό θα πρέπει να το ξαναδούμε. Γιατί να είναι μέλος της πλατφόρμας και να προεδρεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν πολλές, πολλοί λόγοι συντονισμού. Συντονισμό που μπορεί να αναλάβει η Επιτροπή ως προς τον συσχετισμό των διαφόρων δράσεων των Επιτροπών όπου ούτως ή άλλω προεδρεύει η αλλω προεδρευει η Επιτροπή για τη Διοικητική Επιτροπή για, τον, για την κοινωνική ασφάλιση και άλλες επιτροπές, όλες τις επιτροπές που θα πρέπει να συνεργαστούν και να δουλέψουν μαζί για την πλατφόρμα. Επίσης, για να υπάρξει μια συνέχεια στο χρόνο στις δράσεις της πλατφόρμας. Και βεβαίως και η μέρημνα ισορροπία και καλή γνώσης των διάφορων θέσεων των κατόμελων. μελών. Έχουμε διαφορετικές δυνατότητες να συγκεντρώσουμε τις διάφορες επιμέρους γνώσεις μαζί με τις ειδικές γνώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Τέλος για τη μνήα. Στη συγκέντρωση κοινών οικονομικών και τεχνικών πόρων υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως των συστημάτων IT ε, με το πρόγραμμα AEC ή το σύστημα IMI για την ε, εσωτερική αγορά. Αυτές ήταν οι γενικές μου παρατηρήσεις για την ανάγκη αποτελεσματικότητας στην διαχείριση της πλατφόρμας. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ε, Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Περιγινσκή για να πει μια τελευταία κουβέντα, να συνοψίσει. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, ε, ασφαλώς θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για όλους ε, όσους πήραν το λόγο. και που εν γέννη υποστήριξαν τη γενικότερη προσέγγιση της έκθεσης. Και ασφαλώς και για τα πολύ χρήσιμα σχόλια που έκαναν και που σίγουρα θα λεφθούν υπόψη στη μελλοντική μας εργασία. Όντως, ε, είναι μεγάλος ο αριθμός των τροπολογιών που κατατέθηκαν σε ό,τι αφορά και την πρόσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό αποτελεί απόρρια των διαβουλεύσεων κατά τη φάση προπαρασκευής της ε, έκθεσης και φυσικά θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους όσοι με βοήθησαν στην προετοιμασία της έκθεσης γιατί αντιλαμβάνουμε ότι δεν είναι δυνατόν οι προσπάθειε ενός και μόνο ατόμου να αρκέσουν για την προετοιμασία ενό τέτοιου κειμένου. Θα ήθελα να αναφερθώ στα θέματα εκείνα με τη σειρά που τα ακούσαμε του συναδέλφου πριν το λόγο. Να ακολουθήσω λοιπόν μια χρονολογική σειρά. Να ξεκινήσω από το θέμα των ορισμών. Όταν μιλάμε για τη εργασία, τι συζητάμε ακριβώς. Η κυρία Κούνεμα το έθεσε αυτό ιδιαίτερος, αλλά και άλλοι. Και προφανώς εργαζόμαστε με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 1999 ουσιαστικά. Αλλά το εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει τον βασικό ε, νόημα του ότι η αδέλφη εργασία είναι μία απασχόληση επαμοιβή, η οποία δεν είναι στη φύση της παράνομη, δεν είναι εγκληματική δραστηριότητα, ωστόσο δεν καταγράφεται, δεν αναφέρεται στις δημόσιες αρχές και ως εκ τούτου όταν τύφεται το θέμα του τι εννοείται με την νομιμοποίηση, τι εννοείται με την καταγραφή ή αναφορά με απλούς όρους, γιατί η αναφορά σημαίνει ότι για την εν λόγω θέση απασχόλησης θα ισχύει όλο το σύνολο του εργασιακού δικαίου, το καθεστώς κοινωνικών ασφαλίσεων και φοροεπιβολών επιβολών, όπως σε κάθε άλλη θέση εργασίας στο εν λόγω κρατός μέλος. Και εδώ λοιπόν θα αναφερθώ στην προηγούμενη συζήτηση για τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπου αναφέρθηκε ο όρος της ε, συμπερίληψης ως μια βασική προσέγγιση. Μιλάμε λοιπόν για την συμπερίληψη των εργαζομένων στην ε, νόμιμη αγορά εργασίας. Και φυσικά ανακύπτει το ερώτημα του γιατί δεν είναι λοιπόν καταγεγραμμένη αυτή η απασχόληση. Και εδώ θα πρέπει να είμαστε λοιπόν σαφείς, γιατί υπάρχουν ισχυρά δίκτυα που εκμεταλλεύονται τους εργαζομένους και δυστυχώς και επιχειρήσεις, οι οποίες είναι διαδεθειμένες να κάνουν αυτόν τον αθέμητο ανταγωνισμό. Δεν είναι λοιπόν απλό το εγχείρημα του να ρωτήσουμε τον κόσμο και να ζητήσουμε από τον κόσμο να νομιμοποιήσει την θέση απασχόλησής του. Όχι. Είναι θέμα καταπολέμησης των ισχυροτάτων αυτών συμφερόντων. Και όταν ο συνάδελφος μας λέει ότι δεν υπάρχει λόγος να προσπαθήσετε να αναπτύξετε πλατφόρμες και μηχανισμούς στη στιγμή που υπάρχει αυτή η τόσο μεγάλη λιτότητα και πειθαρχία που εξωθεί τον κόσμο στην κατάσταση αυτή, εγώ πιστεύω το αντίθετο. Ακριβώς υπό τις όρους αυτούς, υπό τις συνθήκες αυτές τις τόσο δύσκολες, είναι σημαντικό να μπει ένα τέλος στις πρακτικές τη εργασίας. Φυσικά, κάνοντας ό,τι μπορούμε για να υπάρξει ανάπτυξη, να υπάρξει απασχόληση, να βγούμε από τη λιτότητα, όπως έχει δεσμευτεί η Επιτροπή μας να πράξει αναζητώντας και ευελιξία στο ευρωπαϊκό εξάμεινο, στα διάφορα μέσα, συμπεριλαμβανομένων και όλων των προσπαθειών, να απομακρυνθούμε από τις επισφαλείς θέσεις εργασίας που αναφέρθηκαν και στην προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο και στην ε, ενδιάμεση αναθεώρηση για το 2020. Δύο ειδών θέματα τέθηκαν κατ' ουσία. Καταρχάς ότι πρέπει να υπάρχει μια πιο ισχυρή πλατφόρμα με πιο πολλά δεσμευτικά στοιχεία. Το άλλο θέμα είναι το κατανοητό, η κατανοητή ανησυχία του κατά πόσο να απομακρυνόμαστε από την επικουρικότητα. Μήπως τα κρατημέλη βρεθούν σε μια θέση όπου δεν θέλουν να ακολουθήσουν. Αυτό που θα ήθελα να πω στην παρούσα φάση, Πρόεδρε, είναι ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε το εξή, Να συμπεριληφθούν, να εμπλακούν στην πλατφόρμα αυτή πραγματικά εμπειρογνώμονες. Όχι μόνο επιθεωρητέ εργασία, προφανώς, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και άτομα ιδιαίτερη εμπειρογνωμοσύνης που θα μπορέσουν να κάνουν πολύ συγκεκριμένες ε, προτάσεις και συζητήσεις και όχι μόνο γενικόλογα σχόλια. Αυτό από μόνο του θεωρώ ότι θα μας βάλει σε μια διαδικασία οικοδόμησης εμπιστοσύνης και αυτό τελικά σταδιακά θα μας φέρει πέρα από τη φάση της ανταλλαγής ε, βέλτιστων πρακτικών. Θα μας φέρει στο επίπεδο της ε, κοινή συμφωνία προσεγγίσεων. Να ευχαριστήσω και πάλι τους συναδέλφους και τους κοιόδες εισηγητές, οι οποίοι εξέφρασαν την ελπίδα να καταλήξουμε σε μία κοινή πρόταση με κάποιο βαθμό ευελιξίας και συμβιβασμού χωρίς να χάσουμε την ευκαιρία δημιουργίας ενός ε, φόρουμ όπου μπορεί να επιφέρει ποιοτική αλλαγή στον τομέα αυτό όπου θα συνενωθούν όλα τα κρατημέλη, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, όλοι οι εμπειρογνώμονες και φυσικά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να αναφερθώ στο τελευταίο σημείο τώρα που ανέφερε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά την διακυβέρνηση, τη διαχείριση, πιστεύω ότι το καλύτερο δυνατόν θα ήταν να δοθεί η διακυβέρνηση αυτής του εμπειρογνώμονας των πρωτών μελών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει συντονιστικό, υποστηρικτικό ρόλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Πυρίνσκι, σας ευχαριστώ όλους που συμμετείχατε σε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Χρονοδιάγραμμα ως εξή. Προθεσμία για τροπολογίε 15 Δεκεμβρίου. Έγκριση στην Επιτροπή Επασχόλησης 26 Φεβρουαρίου. Αυτό αποτελεί το στόχο μας. Στην παρούσα φάση μπορεί να αλλάξει φυσικά αυτό. Και τώρα, τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη, αλλά σε καμία περίπτωση το πιο μικρό θέμα τη ημερήσια διάταξη η απαλλαγή. έξι σχέδια γνωμοδοτήσεων για την απαλλαγή για το 2013. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, στην κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλετε μία-μία τις εκθέσεις να σας τις ε, αναλύσω. ό,τι θέλετε, λέει η Πρόεδρος. Ίσως τι το κάνω. Μία-μία και σύντομη, γιατί ξέρω ότι ε, δεν έχουν πάρα πολύ ώρα, δεν ξέρω πώς είναι θα μιλήσουν. Μία-μία καλύτερα, θα είμαι σύντομη. Νομίζω ότι έχουμε μέχρι τις 6.30 λέει η πρόεδρος, αλλά μέχρι τότε θα έχουν φύγει οι συνάδελφοι. Καταλαβαίνω που το πάτε, λέει κυρία Χαρκίνη. Τέλο πάντων, πρώτα απ' όλα, όσον αφορά την, ε, τη γενική απαλλαγή τον προπολογισμών, ε, Βεβαίω και εδώ πέρα είχαμε κάποια, κάποια κάθοδο, κάποια μείωση του ποσοστού φάρματος, στην παράγραφο 3. Ε, εδώ αναφέρονται σε τις παρατηρήσεις του ελεγκτικού συνεδρίου όσον αφορά το σύνομον και εδώ πέρα αναφέρονται τρία πράγματα το ότι έχουμε την επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο, τη διαφοροποίηση των δραστηριότητων και επίσης ε, την πολλαπλότητα των συναλλαγών μικρής και περιορισμένης κλίμακας. Πάρα πολύ σημαντικά για μένα, γιατί εγώ θέλω αυτού του τις συναλλαγές να τις εξετάσουμε σε εθνικό επίπεδο, γιατί οι εκεί συναλλασσόμενοι χρησιμοποιούν τα κοινοτικά ταμεία. Και συνεχώς μου παραπονούνται για την γραφειοκρατία, για τα διοικητικά και δεν είναι καμιά φορά τόσο δύσκολο που δεν ξανά ε, κάνουν τις ενέργειες αυτές να κάνουν αίτηση. Οπότε όπως είπε και το ελληνικό συνέδριο όλα θα πρέπει να είναι βέβαια ε, σύνομα και κανονικά. επίση έχουμε πάρα πολλού ε, ενδιάμεσου σε εθνικό επίπεδο και τα λέει αυτά το ελληνικό συνέδριο. Πάντως θα πρέπει ή δυνατόν να έχουμε κάποιο διάλογο. Αν όχι συνεχή, θα γίνεται δύο-τρεις φορές μεταξύ αυτών των συναλλασσομένων μικρής κλίμακας και της Επιτροπής του Ελεκτικού Συνεδρίου. Και έτσι να υπάρχει κάποιο είδους κατανόηση του πού δυσκολεύει ο μέντον τον δε κλπ. Γιατί οι δυσκολίες που υπάρχουν πέραν των μεγάλων προσπαθειών ότι παραμένουν οι ίδιες δυσκολίες. Αυτό ήθελα να πω. Και κάτι άλλο να πω, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως λέει το συνέδριο, ότι θα πρέπει να υπάρξει τη θέμηνη αξία. Πολλές φορές τα κράτη-μέλη θέλουν να δαπανίσουν τα χρήματα γιατί τα χρήματα υπάρχουν. Επίσης, με μεγάλη μου χαρά διαπίστωσα ότι νέες καθημερινές γραμμές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αναβαθμιστεί η αξιοπιστία κλπ για το περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 θα παρουσιαστεί στα κράτη-μέλη περί τα τέλη ενός φωτός έτους. Οπότε ελπίζω ότι έτσι θα βελτιωθεί η κατάσταση. Και σας ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε εμείς. Πάρα πολύ αποτελεσματικά μας τα είπατε και με σαφήνεια. Για να δούμε τώρα ποιος θέλει το λόγο, κύριος Ρόουλιν. Είσαστε ο σκιώδης εισηγητής για το ΕΛΚΑ λέει ο κύριο Μην επαναλάβουμε ότι είπε η Έχουμε σωστή βάση για να γνωμοδοτήσουμε. Να τονίσω όπως και η συγκήτρια το ότι χρειάζεται διάλογος με τους αλλασσομένους. Γιατί διαπίστωσα και εγώ ότι αυτοί οι μικροσυναλλασσόμενοι έχουν δυσκολίες. δεν μπορούν να ξέρουν πόσα διοικητικά προβλήματα, σε πόσα τέτοια προβλήματα μπορούν να προσκρούσουν για τις αλλαγές τους. Ευχαριστώ. Για τους σοσιαλιστές ο κύριος Πυρίνσκι. Σας ευχαριστώ. Σύμφωνα κι εγώ με τα πράγματα όπως τα είπε η κυρία Χάρκιν. Ήταν εύστοχη να τονίσουμε αυτά που την προβληματίζουν. Μας ε, εξήγησε κάποιο παραδείγματα, Α πούμε στην παραγραφό 3, εδώ πραγματικά πρέπει να τονίσουμε. ότι το ελληνικό συνέδριο προβληματίστηκε με την μη συμμόρφωση των κανόνων για τις δημόσιες κρατικές προμήθειες. Θεωρεί το συνέδριο ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο όσον αφορά τις δράσεις του κοινωνικού ταμείου. Οπότε θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλοι να έχουμε μια πιο ενεργητική στάση. Να αποφεύγουμε τα σφάλματα. μην επεμβαίνουμε μόνο εκ των υστέρων για να διορθώνουμε αυτά τα σφάλματα. Μέχρι το 2013 υπήρξε αυτή η δράση προστασία του υπολογισμού. Εν πάση περιπτώσει, εμείς ε, συμφωνούμε με το κείμενο με την πρόταση. Κύριε Κάρη. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστούμε την συγκεκριά. Άριστα όσο μας είπε. Δεν έχω να πω και πολλά. Συμφωνώ με το σχέδιο κειμένου. Έχει δίκιο για τον διάλογο μεταξύ των συναλλασσομένων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς θα κατεβάσουμε μία-δύο τροπολογίες. Να σας πω γιατί. Τα τελευταία χρόνια είχαμε σημαντικές ενισχύσεις προς τις επιχειρήσεις. Και κάποιες επιχειρήσεις πήραν εργαζομένους, τους προσέλαβαν από άλλο κράτος μέλος. Οπότε αυτοί ως προλογούμενοι συνεισέφεραν σε άλλη χώρα και όχι στην χώρα προελεύσεως τους. Να δει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν αυτό θα συνεχιστεί. Και αυτό είναι, είπαμε, δημιουργία θέσεων απασχόληση, αλλά δεν ωφελεί τη χώρα από την οποία προέρχονται οι σχετικοί εργαζόμενοι. Θέλει κάποιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το λόγο, λέει ο πρόεδρο. Ορίστε κύριε. Ευχαριστώ την κυρία Χάργεν, ευχαριστώ και τους βουλευτές για το σχέδιο Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η γνωμοδότηση αντικατοπτρίζει αυτό που πετύχαμε με την κοινωνική μας πολιτική κλπ. Τα τελευταία χρόνια. Όλα αυτά απορρέουν από την εκτέλεση του προπολογισμού. Αυξήθηκε ο τον πληρωμό το 2014, πήγαμε στα 14 εκατομμύρια και είχαμε συρρήκνωση του ποσοστού σφάλματος. είπαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το gold plating, η απλούστευση. Εμείς έχουμε επενδύσει πολλά σε τέτοιου είδους απλούστευση. Θα συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση. δε περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 είπαμε ότι θέλουμε να έχουμε καλύτερη, περισσότερη απλούστευση. Συνεργαζόμαστε με τα μέρη πάνω σε αυτό. Αυτά έχουμε να σας πούμε και ευχαριστούμε. Πρόεδρος. κυρία Χάρκιν και ίσως και οι οργανισμοί να θέλουν το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα τελικό σχόλιο από αυτόν. Θα ήθελα σε κάποιο σημείο να έχω την ευκαιρία για περαιτέρω συζήτηση και για μια εξήγηση για το πώς ε, λειτουργεί η απλούστευση. Μια λέξη που ακούμε πολύ και στην Επιτροπή Γεωργίας. Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε σίγουροι ότι το πετυχαίνουμε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενο θέμα ο Οργανισμός για την Υγεία και την Ασφάλεια στον Εργασιακό Χώρο. Μερικά σχόλια, όπως και στους άλλους οργανισμούς, το Ελεκτικό Συνέδριο βρήκε ότι είναι νόμιμη και σωστή λογαριασμή και ότι η οικονομική κατάσταση επικονίζεται σωστά. Κάνω δύο σχόλια τώρα, επιτρέψτε μου σε ό,τι αφορά το έργο του οργανισμού και σε ό,τι αφορά τα, τα διαδραστικά εργαλεία με τις μικρομισές επιχειρήσεις για την, ε, ε για την υγεία και την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο και γιατί μιλάμε πολύ συχνά για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις και σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση του πολιετούς ε, σχεδίου. Δεν υπήρξαν ε, μεταφορές απρόβλεπτες. Σημαντικό αυτό γιατί καταδεικνύει ότι τα, οι οργανισμοί προσπαθούν να εφαρμόζουν το πρόγραμμα εργασίας τους. Διορθωτικές δράσεις οι οποίες και συμπεριλήφθησαν, καλώς ορίζονται από το ελεκτικό συνέδριο, σε καλές ε, βελτιώσεις στο τρόπο εργασίας και τρόπο εφαρμογής του ετησίου σχεδίου δράση. και το Μάρτιο συμπεριλήφθησαν δημοσιεύτηκαν προτάσεις. Επίσης, έγινε και ελέγχθηκε η χρήση ενός πειραματικού προϋπολογισμού για το 2013 για το προσωπικό και για διάφορα άλλα έργα. Και πλέον λοιπόν αυτό θα εφαρμοστεί το 2014 για θέματα επίσης πρόσληψης και μισθών του προσωπικού. Και αυτό το θέμα αντιμετωπίστηκε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Σχόλια. Μάλιστα, ωραία. Να πάμε λοιπόν κατευθείαν στο επόμενο θέμα, στον επόμενο οργανισμό για το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ε, επαγγελματική κατάρτιση. Ευχαριστώ. Οι λογαριασμοί είναι όλοι ε, κανονικοί και χωρίς πρόβλημα και με τη σωστή νομική ε, παρουσίαση. Όπως για τον προηγούμενο οργανισμό, κοιτάξαμε το εύστοχο των δράσεων, όπως πρότεινε το συνέδριο, και βάσει των συστάσεων του Κοινοβουλίου. Η δημοσιονομική αρχή του ετήσιου κύκλου, η ενίσχυση του δημοσιονομικού σχεδιασμού, η εξάντε και εξπόστ επαληθεύσεις, και τα δίκτυα των εθνικών συνεργατών και η διαδικασία επιλογής ε, για, δύο, για κάλυψη δύο θέσεων, όλες αυτές οι διαδικασίες θα είναι νόμιμες. Το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω σχετικά είναι ότι το 2014 θα, είναι, θα διεξαχθεί η πρώτη μελέτη, η πανευρωπαϊκή μελέτη για τις επαγγελματικές δεξιότητες. Ειδικώ τώρα που βρισκόμαστε σε περίοδο κρίσης, μερικοί νομίζω δεν καταλαβαίνουν ε, την έλλειψη δεξιοτήτων σωστά. Όταν οι εργοδότες δεν μπορούν να βρουν ε, τους εργαζομένους που αναζητούν με συγκεκριμένε δεξιότητες δηλαδή, τότε μιλάμε για έλλειψη. Είναι άλλο η αναντιστοιχεία δεξιοτήτων. Εκεί μπορεί κάποιοι να έχουν υπερβολικά πολλέ δεξιότητε για θέσει εργασία και αυτό είναι ένα φαινόμενο που διαρκώς διωγγώνεται. Γι' αυτό στην παράγραφο 3 έχω συμπεριλάβει μια πρόταση από ένα έγγραφο που έχει συντάξει το ΣΕΝΤΕΦΟΠ και γι' αυτό είναι σημαντικό να το, σημειώσουμε ότι θα πρέπει να αλλάξει η σύγχρονη τάση για να αντιμετωπιστεί ε, η αναντιστοιχία δεξιοτήτων και η ανεργία. Πιστεύουν κάποιοι ότι αν ε, δώσουμε περισσότερες δεξιότητες στους εργαζομένους θα λύσουμε το πρόβλημα της ανεργίας. Όμως δεν είναι έτσι. Το πρόβλημα είναι πολύ ευρύτερο από την απλή αναντιστοιχία των δεξιότητων με τις θέσεις εργασίας. Yes. Σχόλια. Ναι. Η δουλειά που έγινε εδώ είναι πολύ καλή, όμως πρέπει να τονίσουμε όντως το πόσο καλή δουλειά κάνει το ΣΥΝΤΕΦΟΠ, αλλά μιας και μιλάμε για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και έλεγχο των προϋπολογισμών και για τις ε, ακόλουθες χρονιές, πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι καλύπτονται όλες οι ανάγκες των οργανισμών αυτών και στην προηγούμενη περίπτωση, αλλά και ανάγκες των, των κτηρίων. Ο κύριος Πυρίνσκι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Απλώς να πω ότι είναι σωστές οι προτάσεις της κυρίας Χάρκιν και σωστά αντικατοπτρίζονται και συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Απλώς να τονίσω ότι το ελεγκτικό συνέδριο βρήκε ότι εκθέσεις των οργανισμών αντικατοπτρίζουν τις ε, πραγματικές τους εργασίες και την νομιμότητα των ε, συναλλαγών. Οπότε πρέπει στους οργανισμούς που τώρα εξετάζουμε να αναγνωρίσουμε το σημαντικό τους ρόλο για την εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης και να δώσουμε μια έμφαση στο θέμα των δεξιοτήτων. Νομίζω λοιπόν να προσέξουμε να μην ε, ε, ξεχωρίσουμε κανέναν από τους οργανισμούς που εξετάζουμε αυτή τη στιγμή εις βάρος των υπολείπων. Ευχαριστούμε. Ε, ναι, και τώρα το Ευρωπαϊκό Τρίμα για την επαγγελματική εκπαίδευση. Ναι, και πάλι το ελεκτικό συνέδριο βρήκε ότι οι λογαριασμοί του Ιδρύματος είναι ε, σωστή και νόμιμη και υπάρχει και σωστή ε, παρουσίαση. Η διαρκής συνεισφορά του Ιδρύματος στη δημιουργία τρόπων κεφαλαίου στις χώρες ε, συνεργασίας είναι σημαντική. Αναγνωρίζουμε λοιπόν και αυτού του Ιδρύματος το έργο. Υπήρχε ένα θέμα για το πλεόνασμα του τραπεζικού στα τέλη του 2013, όμως υπάρχει μια απάντηση από το Ίδρυμα που λέει ότι πρώτα απ' όλα το υψηλό τραπεζικό ε, αποτέλεσμα είχε να κάνει με την επιδότηση το 2014 που είχε φτάσει νωρίτερα στους λογαριασμούς για δύο, για τέσσερα μάλλον νέα προγράμματα, το Game και το Frame. Οπότε ήταν απόλυτα λογική η εξήγηση. Ταυτόχρονα συμφωνούμε με τα πορίσματα του συνεδρίου και επιβεβαιώνουν την πρόθεσή τους το 2014 να οργανώσουν κοινή διαδικασία διαγωνισμού για τις τραπεζικές υπηρεσίες που έχει ε, ζητήσει η Επιτροπή και αυτό θα το θίξω και στην τελική γνώμη, την τελευταία από τις γνωμοδοτήσει μου εδώ. Νομίζω είναι σημαντικό να μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους τα Ιδρύματα και οι οργανισμοί. Επίσης για το 99% επίτευξη των επιδόσεων που είχε θέσει ως αρχικό στόχο και για την πρόεδο, πρόοδο που έχει επιτελέσει το Ίδρυμα είναι πολύ θετική η αποτίμηση και για το πρόγραμμα ΠΡΕΜ στις χώρες συνεργασίας. Καταφέρνουν οι διάφορες χώρες να αναλάβουν την ευθύνη για τα προγράμματα και αυτό είναι πολύ σημαντικό βάσει των στοιχείων που λάβαμε. Ήταν πολύ ικανοποιητικά τα αποτελέσματα του Ιδρύματος. Σχόλια. Okay, then we'll go to the... Ωραία. Να πάμε στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθήκων Διαβίωσης και Εργασίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και πάλι σας ευχαριστώ, λέει η κυρία Χάρκιν όλες οι χειρικοί συναλλαγές είναι σύνομες και κανονικές. Πάρα πολύ σωστά παρουσιάζεται η οικονομική θέση του Ιδρύματος τώρα. Όσον αφορά την υπηρεσία αυτή, τόσο στον ότι είχαμε βελτίωση στις περισσότερες επιδόσεις της υπηρεσίας της το 2012, το οποίο είναι θετικό. Επίσης, Είχαμε πολλές μεταφορές πιστώσεων και το συνέδριο έλεγε ότι τα διοτήτα των μεταφορών είχαν προγραμματιστεί το 2014, αλλά επίσης είχαμε και κάποιες εργασίες, 69.000 στον αριθμό, που ήταν εκτάκτου χαρακτήρα και επίσης το 2014 230.000, οπότε έχουμε πάνω από 300.000 τέτοια έξοδα που αφορούσαν και εργασίες ανακαίνησης. Επίσης, είχαμε κάποιο είδους ε, απρόβλεπτες μεταφορές πιστώσεων, ώστε να μπορέσουμε να τονώσουμε την ποιότητα κάποιων προγραμμάτων, ε, μεταφραστικές υπηρεσίες, μέχρι Δεκέμβριο του 2013, αλλά αυτό είχε προγραμματιστεί το 2014, ε, επίσης σε σχέση με τις προμήθειες είχαμε κάποιους και από πλευρά των αντισυμβαλλωμένων αλλά νιώθηκαν απειμένοι από τις ε, παρασχεθήσει εξηγήσει. Δεν ξέρω αν κάποιο έχει κάποια ένσταση. Εγώ νομίζω ότι όλα αυτά είναι σύνομα και κανονικά. Επίσης, επίσης είχαμε πέρυσι την αναγνώριση του πόσο το Eurofound προσφέρει ποιοτικέ επιστημονικές εργασίες, να κοιτάξετε τις ε, ε, δημοσιεύσεις, επιστημονικά ε, περιοδικά κλπ. Οπότε όλα αυτά καταδεικνύουν ότι έχουμε εδώ πέρα ψηλή ποιότητα υπηρεσίες που προσφέρει αυτό το Ίδρυμα. Έχετε παρατηρήσεις, λέει η Πρόεδρος. Κύριε Πυρίνσκι. Δύο λόγια μόνο όσον αφορά αυτή την υπηρεσία. Ίσως οι συνάδελφοι έχουν παρατηρήσει ότι πρόκειται για την υπηρεσία στην οποία θα στηριχθούμε πάρα πολύ για την πλατφόρμα την οποία συζητήσαμε. Έτσι θα έχουμε μία τράπεζα, μία αποθήκη γνώσεων Ήδη είναι, είναι εντυπωσιακές οι επιδόσεις αυτής της υπηρεσίας. Επομένως, αυτό το οποίο επιβάλλεται είναι να παρακολουθούμε προσεκτικά πώς δαπανούνται οι πόροι για αυτό το ίδρυμα. Επίσης, νομίζω ότι ε, οι φιλόδοξοι στόχοι του Ιδρύματος αξίζουν της υποστήριξής μας. Πρόεδρος. Θέλω να πάμε στην τελευταία υπηρεσία. Α, όχι, κύριε Ρολά, έχει πει το λόγο. Συμφωνώ 100% με τις ε, προτάσεις και να τονίσουμε το πόσο σημαντικό είναι το έργο της υπηρεσίας αυτής το Διεθνές Γραφείο εργασία, να ξέρετε ότι αναφέρεται συνεχώς στο έργο της υπηρεσία την οποία συζητούμε. Σας ευχαριστώ λέει Τώρα, κύριε Χάρκιν, τελευταία έκθεση όσον αφορά την εκτέλεση του προπολογισμού για τη χρήση 2013 όσον αφορά αυτές τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Κύριε Χάρκιν, σας ευχαριστώ. Όπως είπαν οι συνάδελφοι, έχει βοηθήσει η υπηρεσία αυτή, η υπηρεσία για τη βελτίωση των συνθήκων ε, διαβιώσεως και εργασίας. Βοηθά και για την ε, στρατηγική των στόχων 2020. Ε, Επίσης, είναι σημαντικό και τους στόχους του 2020, τα προγράμματα και οι στρατηγικές να αντικατοπτρίζουν τις υπάρχουσες προτεραιότητες. Να είμαστε συνεπείς δηλαδή προς τις προτεραιότητες που έχουμε τάξει. Παράγραφοι 3 και 4 αλλά και οι 5 αναφέρονται στο χαρτιπορία στην κοινή προσέγγιση Υπήρξε μια τέτοια που συνεφωνήθη το 2012 τον ε, Ιούλιο. Συμφώνησαν τα τρία θεσμικά όργανα. Το δε, Δεκέμβριο, πριν από δύο χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι θα κάνει το χαρτί πορείας σε συνέχεια της προσεγγής εκείνης. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό με ε, συντομία να δούμε τι προβλέπει ο χαρτής πορείας και πού πηγαίνουμε με αυτόν. Επίσης θα πρέπει να τονίσουμε και κάποια άλλα σημεία. Ας πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει κάποιες αντιθετικές γραμμές για κάποιες συμφωνίες. Κάποιες από αυτές τις έχουμε συζητήσει, όχι όλες όμως. Ο χάρτης πορείας αυτός επίσης εξορθολογίζει τη λειτουργία των ε, υπηρεσιών αυτών. Ας πούμε, η υπηρεσία της Λισαβόνας για την καταθαλασσά ασφάλεια είπαμε ότι ε, τώρα ε, συνδέθηκε με την υπηρεσία του Βίγκο έκανε συμφωνία τέλος πάντων και η υπηρεσία επίσης των σιδηροδρόμων επίσης ε, συμφώνησε για την υπηρεσία θαλάσσιας πολιτικής σε σχέση με κάποιον όνοτρο αξιωματούχο. Αυτά εννοεί η παράγραφος 3 και αναφέρει την ε, Europol επίσης. Έχουμε επίσης ένα χειρίδιο για την ευθυντική γραμμή για τις υπηρεσίες αυτές. Επίσης βλέπουμε για τον προγραμματισμό, τον πολιετή, αλλά και τον ετήσιο και τη σχετική έκθεση. Επίσης, τι γίνεται για την ε, άρση, την επίλυση διαφορών σύγκρουσης συμφερόντων. Είναι κάποια σημεία που αφορούν όλες τις ε, υπηρεσίες. Επίσης, θα δούμε τι γίνεται όσον αφορά τον κανονισμό για το δημοσιονομικό, χρηματοδοτικό πλαίσιο, οι υπηρεσίες, streamlining, για την, για την ένταξη πολιτικών στις ε, στο έργο του, του έργου του στις πολιτικές μάλλον, επίσης ε, χρηματοδότηση πολιετών ε, προγραμμάτων και έχουμε τώρα κάποιους δείκτες επιδόσεων τους οποίους επεξεργαζόμαστε για να δούμε πώς πάνε οι επιδόσεις τους και αυτά όλα έχουν ζητηθεί με τις ε, αποκεντρωμένες αυτές τις υπηρεσίες. Από ό,τι ξέρω όμως δεν έχει αποκρισταλωθεί μια θέση. Όλα αυτά είναι βήματα τα οποία έχουν ληφθεί στα πλαίσια του χαρτιπορίας για να μπορέσουμε να ε, βελτιώσουμε την λειτουργία αυτών των υπηρεσιών και να έχουμε ένα συνεπές λογικό λειτουργικό πλαίσιο. Εμείς θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε έχουμε παρατηρήσεις. Ε, επιτρέψτε μου να σημειώσω ένα-δυο στοιχεία αναπτύσσοντας την τόσο καλή βάση που μας προσέφερε η κυρία Χάρκιν για τις κατευθυντήριες γραμμές και τις βασικές διατάξεις για τη συμφωνία Για τα γραφεία των αποκεντρωμένων οργανισμών, από το 2 βλέπουμε ένα, τρίτο των 32 αποκεντρωμένων οργανισμών να μην έχουν εφαρμόσει πλήρως την ε, συμφωνία για τα κεντρικά γραφεία. Αυτό ε, έχει να κάνει βεβαίως και με τους όρους που έχουν πετύχει για τα κεντρικά γραφεία και τον να υπάρχουν ελκυστικοί και διαφανείς στη λειτουργία του χώροι. Ως προς τι επιδόσει, των σχεδιασμών προπολογισμού, ε, καλό είναι να τονίσουμε εδώ την ανάγκη ευθυγραμμισμού του συντονισμού και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Κατευθυντήριες ε, γραμμές για την ε, στρατηγική των οργανισμών ως προς την καταπολέμηση της απάτης, όπως προτείνει και η όλα. Δύο εργαστήρια έπρεπε να έχουν διεξαχθεί το 2014. Και επειδή έγινε αυτό, υπήρξε και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Βάσει των όσων είπε λοιπόν υπέρ ε, του εξορθολογισμού, των template και των κατευθυντήριων γραμμών για τους οργανισμούς, νομίζω ότι με όλα αυτά θα βελτιωθεί η λειτουργία των ε, ε, οργανισμών αυτών. Ο κύριος Γολά, να προσθέσω για το σημείο 4 και τις προσπάθειες που απαιτούνται για τον εξορθολογισμό, ότι και καταλαβαίνουμε και στηρίζουμε αυτή την προσέγγιση, αλλά εκτός από το ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ως προς το έργο των οργανισμών και των ιδρυμάτων, εκτός από τους τριμερείς οργανισμούς, θα πρέπει να βεβαιωθούμε για τον δυναμικό χαρακτήρα και την ποιότητα της δουλειάς που κάνουν. Ευχαριστούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να πει κάτι. Παρακαλώ. Πολύ σύντομα να πω ότι συμφωνούμε με τις πληροφορίες και την αξιολόγηση που έγινε εδώ για την εφαρμογή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιας κοινή προσέγγισης από το 2011 ο δικός χάρτης που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2012 ε, περιλαμβάνει 90 μέτρα. Δεν πρέπει όλα να τα φέρει πέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε μερικέ περιπτώσει τα ιδρύματα και οργανισμοί να αναλάβουν, αλλά υπάρχει όντω πρόοδο ως προς την εφαρμογή του δικού χάρτη. Ιδίω ω μια πτυχή που πρέπει να τονιστεί. Μεταξύ των μέτρων αυτών αναφέρεται και η ανάγκη αναθεώρησης των ιδρυτικών κανονισμών σε ορισμένες περιπτώσεις. Ιδίως όταν αυτοί είναι απαρχαιωμένοι και δεν συμπεριλαμβάνουν τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την διαχείριση και βάσει των συστάσεων της κοινή προσέγγισης. Αυτή την νομοθετική δουλειά ε, την έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήδη έχουν προταθεί κάποιε αναθεωρήσει. Κάποιε άλλε ακόμη μελετώνται, ιδίω για να τι συμπεριλάβουμε στο πρόγραμμα εργασία του 2015. Ευχαριστούμε. Άρα, ολοκληρώσατε κυρία Χάρκιν. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Ε, το χρονοδιάγραμμα, η προθεσμία μάλλον, η λήξη της προθεσμίας για την υποβολή τροπολογιών είναι 9 Δεκεμβρίου και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 29 Ιανουαρίου. Αυτό σημαίνει ότι ε, λίγη συνεδρίαση, αλλά, αλλά οι συντονιστές ελπίζω να μείνετε. Να μείνετε γιατί έχουμε αναγγείλει συνεδριές των συντονιστών. Θα είναι πολύ γρήγορη, θα ξεκινήσει στι 6, οπότε θα έχετε ένα μικρό διάλειμμα, ένα intermedio. Και θα ζητήσω και από τους διερμηνείς εάν μπορούν να μείνουν ως την πολύ σύντομη συνεδρίαση συντονιστών μας στις 6. That is possible. Yes. Thank you very much.